Good afternoon, everybody. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ, καθίστε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι δυόμιση το απόγευμα. Συνήθως ξεκινάνε οι συνεδριάσεις στις 3 το απόγευμα. Οπότε ενδεχομένω κάποιοι συνάδελφοι θα έρθουν στην πορεία. Έχουμε όμως μία ώρα να αφιερώσουμε σε αυτή τη συζήτηση για να τηρήσουμε και το πρόγραμμά μας. Έχουμε εδώ στο πρώτο σημείο τη απογευματινή συνεδρίαση κοινή συζήτηση με τρει επιτροπέ. Την Επιτροπή Ανάπτυξη, την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη δική μα φυσικά, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχω εδώ στα αριστερά μου τον κύριο Ντάνιελ Έντρε, που είναι διευθυντή ΥΠΑ τη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο Φόρουμ για του Πρόσφυγε. Και να σα ενημερώσω λίγο για το υπόβαθρο και προ τι αυτή η κοινή συζήτηση των τριών επιτροπών. Επίκειται το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για του Πρόσφυγε που θα λάβει η χώρα 15 με 18 Δεκεμβρίου 2019 στη Γενέβη. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για το Άσυλο υιοθετήθηκαν το 2018 από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εξού και αυτό το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους πρόσφυγες θα είναι ευκαιρία για να αναγγελθούν συγκεκριμένες υποσχέσεις και συνεισφορές από διαφόρους εμπλεκομένους, παρουσία κρατών μελών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε έναν επιμερισμό του άχθους και της ευθύνης μεγαλύτερο από ό,τι μέχρι τώρα. Και περιμένουμε την παρουσίαση του εκπροσώπου της ΥΠΑ της Αρμοστίας, του κυρίου Ντάνιελ Έντρες, που θα τροφοδοτήσει και τις δικές μας συζητήσεις και θα μας βοηθήσει στην προετοιμασία της ad hoc μας ε, αντιπροσωπείας το Δεκέμβριο στη Γενέβη. Και μάλιστα πριν από μία ώρα είχαμε και προπαρασκευαστική συνεδρίαση και εκεί είχαμε ήδη μια προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Αντρές, αλλά η ανταλλαγή αυτή απόψεων θα συνεχιστεί τώρα στη δημόσια συζήτηση παρουσία των τριών επιτροπών. Δεν ξέρω αν η κυρία Ρενά ή κάποιος άλλος ήθελαν το λόγο και μετά θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά αγαπητέ πρόεδρε και να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την πρωτοβουλία αυτή της ε, συντονιστικής προπαρασκευαστικής ε, συνάντηση με τον Αντρές, παρουσία των τριών επιτροπών που είναι αρμόδιες για το θέμα αυτό. Και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα δόθηκε το ανακτήριο λάκτισμα στη Νέα Υόρκη για το σύμφωνο, Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε συναρμόδιες τρεις ε, επιτροπές και θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία συνεχή και σοβαρή παρακολούθηση των ε, τριών μηχανισμών. Έχουμε τη συζήτηση στην ε, Γενική Συνέλευση, ε, τις διερευνητικές επιτροπές, αλλά και τον Απρίλιο είχαμε σχετικό ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα έχουμε μια μελή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρτίζεται από μέλη των τριών επιτροπών και ήδη συμμετείχαμε στην διακυβερνητική διάσκεψη για, στο Μαρακές 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018 για την υιοθέτηση του Παγκοσμίου Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Έτσι, με την ad αυτή την προσωπία, θα έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη ε, θεώρηση και εξασφάλιση της συνέχισης του έργου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς ως συνομοθέτες ε, του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού θα πρέπει να συμβάλλουμε στην εφαρμογή των δύο αυτών παγκοσμίων συμφώνων, ώστε ε, να γίνονται σεβασμό, σεβαστά το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο για τις αναγκαστικές μετακίνησει, το άσυλο και τη βοήθεια των κοινοτήτων ή χωρών υποδοχής. Χαίρομαι εκ των προτέρων για αυτή τη συνεργασία που θα καλύπτει την εσωτερική διάσταση του δικαίου αλλά και την εξωτερική διάσταση αυτής της μείζωνος πρόκλησης των καιρών μας με σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων. Ο κύριος Τόμπε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συμπρόεδροι και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να τονίσω τη σημασία που έχει αυτή η εκδήλωση και πόσο στην, στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, ενδιαφερόμαστε για αυτό το θέμα των αναγκαστικών μετακινήσεων που έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδο τα τελευταία χρόνια. 17,8 εκατομμύρια άνθρωποι ε, μετακινήθηκαν αναγκαστικά ανά τον κόσμο. 87% αυτών των ε, προσφύγων διαμένουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και 26 χρόνια είναι η διάρκεια που περνάει κάποιος σε αυτή τη ε, μετατόπιση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τις κοινότητες και υποδοχής και να εξασφαλίσουμε την ε, επιστροφή στις αιστείες τους ή την επανεκατάσταση. Οι πρόσφυγες δεν μπορούν να εξαρτώνται για γενιές ολόκληρες από βοήθεια εξωτερική. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε ε, επαρκώς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής και η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να επιτρέψει τους πρόσφυγες και ε, μετανάστες να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και να έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες, ε, στην αγορά εργασίας, ε, στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε και τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Αντρές. Θα έχουμε όμως στη συνέχεια χρόνο για συζήτηση, οπότε όποιος θέλει το λόγο μετά να το δηλώσει τώρα ή αργότερα, δίνοντας το όνομά του ή σηκώνοντας την κάρτα του. Και ίσως θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για να μας πούν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο και το αντικείμενο αυτού του Παγκόσμιου Φόρουμ για τους πρόσφυγες που θα γίνει το Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και αξιότιμοι βουλευτές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να συζητήσω το Παγκόσμιο Φόρμιο της Πρόσφυγες μαζί σας ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα και τα κρατημέλη αποτελούν εταίρο, σταθερό σε ό,τι αφορά αυτή την πολυμερή διεθνή τάξη. Ένα χρόνο μετά την ε, έγκριση του Παγκόσμια Συμφωνίας για τους πρόσφυγες, βλέπουμε πλέον να διαγράφεται η ευκαιρία να μεταγραφεί, να μετατραπεί αυτό το σύμφωνο σε πραγματικότητα με το Παγκόσμιο Φόρουμ Προσφύγων που θα λάβει η χώρα, όπως είπε ο πρόεδρο στι 16 έως 18 Δεκεμβρίου στη Γενέβη τη Ελβετία. Η επίλυση της κατάστασης των προσφύγων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διεθνούς συνεργασίας. Και εμείς, ε, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, προσβλέπουμε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το σύμφωνο για τους πρόσφυγες. Τρία θέματα θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς θα ήθελα να μιλήσω για το περιεχόμενο συγκεκριμένα του φόρου. Στη συνέχεια θα ήθελα να επικεντρωθώ στο τι θέλουμε να πετύχουμε και στο τρίτο τμήμα της παρουσίασης μου θα ήθελα να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα για να μετατραπεί, να υλοποιηθεί αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο. Το σύμφωνο λοιπόν άλλαξε τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος σε καταστάσεις που αφορούν πρόσφυγες. Μεταφράζει την ιδέα της διεθνούς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένες δράσεις. Δράσεις για πιο σωστή, ίση κατανομή των του άχθου σε ό,τι αφορά του πρόσφυγε. Αν κοιτάξουμε τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2020, τι έγινε. Ο κόσμο έχει δει να ξεσπούν νέε κρίσει. Συρία, Βενεζουέλα, Ουκρανία. Ενώ καμία από τις παλιέ διαμάχες δεν έχει επιληθεί ουσιαστικά. Άρα αυτά τα 10 χρόνια ο αριθμός των εκτοπισμένων ανθρώπων έχει διπλασιαστεί. Και όπω είπατε και εισαγωγικά, Είμαστε πλέον ε, περίπου στα 71 εκατομμύρια άτομα τα οποία είναι εκτοπισμένα. Επίσης, 85% των ε, εκτοπισμένων ζουν στις πιο φτωχές χώρες του κόσμου και έχουν πολύ α, ανεπαρκή υποστήριξη ακόμα και τώρα. Και επειδή οι πρόσφυγες επιγενιές παραμένουν σε κλειστά καταλήγματα για πρόσφυγες, περιμένουν συζήτεια Αυτή η κατάσταση λοιπόν κρίνεται εντελώ ανεπαρκή και γι' αυτό λοιπόν το σύμφωνο για του πρόσφυγε ζητά μια ριζική αλλαγή προκειμένου να συμπεριληφθούν οι πρόσφυγε στι ε, τοπικέ κοινωνίε και να υποστηριχθούν αυτέ οι κοινότητε με ανθρωπιστική ενίσχυση και με μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις ε, στον δυτικό κλάδο, όπως αναφέρθηκε. Το Παγκόσμιο Φόρουμ για του Πρόσφυγες, λοιπόν, θέλει να καταστήσει λειτουργικό το Παγκόσμιο Σύμφωνο και να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα να δραστηριοποιηθεί πιο πολύ και καλύτερα για τους πρόσφυγες αυτού τι κοινότητε αυτές. Το Παγκόσμιο Φόρουμ θα, λάβει χώρα, θα λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια σε υπουργικό επίπεδο και θα έχει πολλού εμπλεκόμενου φορεί για να είναι πιο ευρεία η υποστήριξη προ του πρόσφυγε. Θα συνενώσει λοιπόν, θα συγκεράσει κυβερνήσει, τοπικέ ε, και περιφερειακέ ενώσει όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τον ιδιωτικό κλάδο, τον ΟΗΕ, τον ακαδημαϊκού κύκλου, ε, την κοινωνία των πολιτών, τι κοινωνίε υποδοχή και φυσικά του ίδιου του πρόσφυγε. Το πρώτο φόρουμ θα λάβει χώρα, όπω είπαμε, το Δεκέμβριο και ο ΙΕ και η Ελβετία συνδιοργανώνουν το φόρουμ αυτό. Πέντε κρατημέλη επίσης έχουν αναλάβει την ηγεσία, είναι υπό την αιγίδα τους λοιπόν το φόρουμ αυτό, μαζί με την ΟΗΕ, η Κωνσταντίνα, Αιθιοπία, Πακιστάν και Τουρκία. Τα κρατη λοιπόν αυτά θα εκπροσωπούνται από τον αρχηγό κρατών και κυβερνήσεις. Στα διάρκεια του φόρουμ, οι ηγέτε και οι άλλοι φορείς θα έχουν ε, την ευκαιρία να καταγράψουν τα όσα έχουν λάβει η χώρα, να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές και το πιο σημαντικό ασφαλώς, να ανακοινώσουν συγκεκριμένε δεσμεύσεις και νέα βήματα τα οποία θα κάνουν για να υποστηρίξουν του τέσσερις ευρύτερου στόχου του συμφώνου, οι οποίοι είναι οι εξή. Καταρχάς, να απαλύνουμε την πίεση στις χώρες υποδοχή, όπως είπαμε ήδη, ιδιαίτερα στις ε, χώρες πυρήνα, η οποία, ή, στις χώρες τη πιο που δεν υποστηρίζονται σωστά. Δεύτερο στόχο, να βελτιωθεί το καθεστώ ε, αυτάρκειας των προσφύγων. Οι πρόσφυγες που περιμένουν γενναία επί γενναίων σε ε, καταβλισμούς χρειάζονται πρόσβαση στην κοινωνία, χρειάζονται πρόσβαση στην εκπαίδευση για να μπορέσουν και αυτοί να συμβάλλουν με την εργασία τους. Και να είναι προς όφελος αυτό προφανώς όλου του κράτους. Τρίτος στόχος, προφανώς να υπάρξουν λύσεις που να ενέχουν και τρίτες χώρες, επανεκατάσταση για παράδειγμα. Και τέταρτος στόχος, να υποστηριχθούν ή να βελτιωθούν οι συνθήκες στο κράτος προέλευσης, ώστε οι πρόσφυγε να μπορέσουν να επιστρέψουν στι χώρε του, ελπίζουμε με καλύτερα εφόδια και με καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση. Σε αυτό το φόρουμ, λοιπόν, έξι είναι οι τομεί οι οποίοι εντοπίστηκαν ω τομεί ιδιαίτερη προτεραιότητα. που επίσης υποστηρίζονται από τα κράτη-μέλη κλειδί και με χαρά αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ε, κατανομή των βαρών, θέσεις απασχόλησης ε, και πολλούς άλλους στόχους. Ε. Σε ό,τι αφορά το, την κατανομή του άχθους. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη διεθνή συνεργασία, να υπάρχει καλύτερη αλληλεγγύη στις κοινότητες υποδοχής, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση μαζί με τους πρόσφυγες. Κατά δεύτερον, η εκπαίδευση. Όπως τα ξέρετε, οι μισοί σε όλο τον κόσμο είναι παιδιά και παρόλα αυτά 4 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτό καθιστά τους πρόσφυγες ε, την ομάδα του πληθυσμού που έχουν μείνει πιο πολύ πίσω από κάθε άλλη σε ό,τι αφορά την παιδεία. Πώς λοιπόν να οικοδομήσουμε το μέλλον μας χωρίς ε, εκπαίδευση. Τρίτος κλάδος, η θέση της απασχόλησης και πόσο σημαντικό είναι να ενταχθεί και αυτό στο πρόγραμμα. Είναι προφανές. Τέταρτη ομάδα, ενέργεια και υποδομές. Καθαρή ενέργεια προφανώς. Και να μην ξεχνάμε ότι όσο έχει η κατάσταση με τους ε, πρόσφυγες, με 40% των πρόσφυγων να μένουν σε καταβλισμούς, στους οποίους καίγονται καθημερινά 500 τόνοι ξύλου για θέρμανση και για μαγείρεμα. Υπάρχουν πιο οικολογικοί τρόποι. Και τέλος, ε, προστασία και εξεύρεση λύσεων. Πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν με καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των προσφύγων. Τώρα, θα ήθελα στο δεύτερο σημείο αυτό να συνοψίσω τα βασικά πορίσματα, τα, τα βασικά αποτελέσματα στα οποία προσβλέπουμε, τα οποία προσδοκούμε. Έχω δέκα σημεία σας τα οποία σας τα έχω μοιράσει. Αν δεν τα έχουμε εδώ πέρα, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Θα μιλήσω μόνο για δύο-τρία εξ αυτών. Το πρώτο θέμα. Πώς μπορούμε να διευρύνουμε τη βάση της υποστήριξης. Αν κοιτάξουμε τις, τα 193 μέλη του ΟΗΕ, 40-50 μόλις είναι σοβαροί δωρητέ οι χώρε υποδοχή για την υποστήριξη των προσφύγων. Έχουμε μια μεγάλη λοιπόν ευκαιρία να τη βρίνουμε τη βάση αριθμητικά σε ό,τι αφορά τις χώρες που είτε είναι χώρες υποτοχής, είτε δραστηριοποιούνται σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό κλάδο, τομέα. Δεύτερο αποτέλεσμα στο οποίο προσδοκούμε. Οι χώρες υποδοχής να συμπεριλάβουν τους πρόσφυγες στα σχέδια ανάπτυξης, γιατί μόνο στην περίπτωση αυτή θα είναι δυνατόν να μπορέσουν οι πρόσφυγες πραγματικά να πάνε σχολείο, να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η υποδομή να λάβει υπόψη και την αύξηση προφανώς του πληθυσμού. Θα ήθελα αυτά να τα συνδέσω με το τέταρτο ευκταίο αποτέλεσμα. Οι πρόσφυγες να μην υποστηρίζονται μόνο από ανθρωπιστική άποψη όπως γίνεται στην παρούσα φάση. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είμαστε ευγνώμονε προς την ΕΚΟ, ένα από τους μεγαλύτερους δωρητέ μας, ε, που όχι μόνο μα δίνει χρηματοδότηση, αλλά και προστασία. Οι πρόσφυγε θα πρέπει να συγκαταλέγονται στου ε, παράγοντες που λαμβάνουν αποφάσεις, ακριβώς επειδή παίρνει τόσο πολύ καιρό η λήψη αποφάσεων. Και εδώ βλέπουμε να τα πιστρεοποιείται η ΔΕΦΚΟ και άλλοι φορείς της ευρωπαϊκή Ένωσης για να μπορέσουν να τη βρίνουν τη βάση αυτή στις χώρες και εδώ σημαντικό ρόλο παίζει και η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία έχει ειδικό παράθυρο αφιερωμένο στους πρόσφυγες 200 δις ευρώ, δολάρια, συγγνώμη, ε, υπό το πρόγραμμα AIDA προς την παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες. Να έρθω τώρα στο τρίτο θέμα, στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παρέμβει με τρόπο συντονισμένο στο φόρουμ για να προωθήσει το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Ειδικά το Κοινοβούλιο μέσω των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του και ως βασικό εποπτικό θεσμικό όργανο είναι απολύτως απαραίτητο για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους ε, πρόσφυγες σε σχέση με τον θεσμικό σας ρόλο η Πατερμοστία αναμένει διαβουλεύσεις για το νέο σύμφωνο αυτό, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ και αναμένουμε από το Κοινοβούλιο και το Συμβουλίο να μεταρρυθμίσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έτσι ώστε να αυξηθεί ο χώρος προστασίας στην Ένωση και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την δική μας στήριξη στην διαδικασία αυτή. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πολλά να επιδείξει. Πρώτα απ' όλα θα τόνιζα την σημαντική πολιτική για τις ε, ζωές και την αξιοπρέπεια κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον προσφυγικό κόσμο και επηρεάζει επίσης και αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα στο σχετικό σύμφωνο. Δεύτερον, Εκτιμούμε επίσης ε, την αυξημένη χρηματική στήριξη στις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες. Εκεί πέρα έχει κάνει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι πρέπει με το νέο ΠΔΠ να δείτε πώς αυτό μπορεί να γίνει με πιο θεσμικό και συστηματικό τρόπο και επίσης να τονίσω την ε, σημασία εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιφερειακές διαδικασίες όπως το κέρας της Αφρικής για ζητήματα συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρμαχος της πολυμέρειας και ο μεγαλύτερος πάροχος βοηθείας παγκοσμίω. Και έχει πάρα πολλά μέσα στην διάθεσή της ε, για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Ε, το ιδεώδες θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να κινητοποιεί περαιτέρω χρηματοδότηση πέρα από την τακτική αναπτυξιακή βοήθεια μέσω δίμερων και πολυμερών διάβλων με άμεσα ωφέλη για τις ε, χώρες υποδοχής και τους πρόσφυγες. Μόνο αν γίνει αυτό θα δούμε έναν αντίκτυπο στις χώρες που χρειάζονται ένα επιπλέον κίνητρο. Επίσης, απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει το επόμενο πολίτες πλαίσιο, ειδικά το μέσο γειτονία για να αυξηθεί η ανθρωπιστική χρηματοδότηση και να συνεισφέρει στις κοινότητες που φιλοξενούν. Επίσης, απευθύνουμε έκκληση στην ένταξη των προσφύγων στις μεγάλες χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει την αναπτυξιακή της βοήθεια σε περιπτώσεις εκτοπισμένων και να έχει αποκλειστική χρηματοδότηση για να προλάβει αυτά τα ζητήματα και να τα αντιμετωπίσει. Η επιπλέον χρηματοδότηση μπορεί να προλάβει την περαιτέρω μετακίνηση και να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι πιο κοντά στα σπίτια τους όπου θέλουν να είναι έτσι ώστε να μην απληπίζονται και να κάνουν επικίνδυνα ταξίδια για να φτάσουν την Ευρώπη ή άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά η χρηματοδότηση από μόνη της θα έχει πραγματικό αντίκτυπο μόνο εάν συνοδευτεί από αλλαγή πολιτικής. Η πρόσφατη εμπλοκή της Παγκόσμιας Τράπεζας, ε, με συγχωρείτε κύριε Έντρες, μιλάτε ήδη 15 λεπτά και έχουμε κάποιους βουλευτές που θα ήθελα να πούν και αυτοί κάποια πράγματα. Αν μπορείτε λοιπόν συντομεύετε, γιατί βλέπω ότι έχετε ακόμα κάποιες σελίδες. Όχι πολλές, μάλιστα. Πάνω στην ώρα κύριε Πρόεδρε, γιατί ολοκληρώνω. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ βασικό σημείο όμως. Να τονίσω πως η ευρωπαϊκή διπλωματία βεβαίω με στον αντιπροσωπιών της Ένωσης και με όλα τις, ε, τα μέσα παίζει ρόλο κλειδί στο να αντιμετωπίσει τις και στην επίλυση των συγκρούσεων. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας το εξής. Μέχρι τώρα βοηθούσαμε τους προσφύγες να επιζήσουν. Με το σύμφωνο πρέπει να τους δώσουμε ένα μέλλον και για τις ε, κοινότητες που τους υποδέχονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ικανότερο θεσμικό όργανο για να κάνει κάτι τέτοιο και ζητώ συγγνώμη που ξεπέρασα τον χρόνο κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι βέβαια, σωρές. Είστε προσκεκλημένος και ευπρόσδεκτος. Ε, βεβαίως οι ανισχύες της ΥΠΑ της ε, του ΟΗΕ ήταν πάντα παρούσες στην συζήτηση της Επιτροπής μας αυτά τα οποία αναφέρεται ειδικά για την ανάγκη νομίμων διόδων για να καταργήσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο της παράνομης ε, διακίνησης και να έχουμε μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση. Όλα αυτά ε, πάντα ήταν ουσιαστικά για την πλειοψία της Επιτροπής μας, τουλάχιστον στην Επιτροπή μας, ε, να είστε σίγουρος. Να σας πω ότι υπάρχει και μία αντιπροσωπεία προς το φόρουμ αυτό των προσφύγων που αποτελείται από εννέα βουλευτές των ε, τριών επιτροπών. Θα προεδρεύω εγώ, θα υπάρχει η κυρία Γουόλς, ε, η κυρία Σιλβάνα, Φονβίζε, Τσίμιοκ, και η κυρία Μαλμπιόρκ. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περιλαμβάνεται στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τούτου λεχθέντος, γιατί τα ξέρετε αυτά, γιατί είχαμε και την προπαρασκευαστική συνεδρίαση. Ε, ας δώσουμε τον λόγο στους συναδέλφους. Βεβαίω ε, έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε στον προσκεκλημένο μας τα μέλη της αντιπροσωπείας που ανέφερα θέλουν να μιλήσουν. Μετά οι υπόλοιποι, τους σημείωσα, η κυρία Μπιόρκ και κάποια άλλη. Θέλουν να μιλήσετε. Κύριος Κάρεμ. Να ξεκινήσετε εσείς, κυρία Μπιόρκ, μια που θα προεδρεύετε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον κύριο Έντρε που ήρθε στην Επιτροπή και ευχαριστούμε και για τις φιλοφρονήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιτεύγματά της. Μερικοί από εμά, ξέρετε, ήμασταν αρκετά επικριτικοί για τις αδυναμίες και για το τι δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε. Προσβλέπω στη συμμετοχή μου σε αυτό το φόρουμ, το περιμένω με ανυπομονησία και πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπου και εκεί για να αυξήσουμε την ικανότητα προστασία των προσφύγων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι η στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ε, ε, επανεγκατάσταση, που είναι ένας τρόπος εξασφάλιση προστασίας. Πάντως, μερικοί είναι κατά ε, της αυθόρμητης άφηξη. Ε, και αίτηση σύλλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που δικαιούνται κάτι τέτοιο με βάση τη συνθήκη τη ε, Γενέβη. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, ούτε είναι αντιφατικά αυτά. Θα πρέπει αυτό να αποσαφινιστεί ε, στη συνεισφορά μα στο Παγκόσμιο Φόρουμ για του πρόσφυγε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αύξηση τη ικανότητα προστασία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Χαιρετίζω την πολυμερή προσέγγιση. Χαίρομαι που η πολυμέρεια θα χαρακτηρίσει αυτό το φόρουμ. Θέλουμε στενή συνεργασία με τι κοινότητε προσφύγων και με τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντε στην όλη διαδικασία και χωρί τη βοήθεια των ΜΚΟ δεν πρόκειται να δώσουμε μια ουσιαστική λύση στο θέμα αυτό. Και επαναλαμβάνω, προσβλέπω και στη συζήτηση που θα έχουμε επί της εκθέσεώς μου στην Αρμόδια Επιτροπή. Είχαμε αρκετά επιτεύγματα σε ό,τι αφορά τα σχέδια επανεγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο και περισσότερε χώρε συμμετέχουν. Αλλά ανησυχώ γιατί δεν έχουμε ε, μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι περισσότερο ad hoc οι δεσμεύσεις, είναι υποσχέσεις που αναλαμβάνονται ετησίως. Θέλουμε κάτι πιο βιώσιμο, πιο μακροπρόθεσμο, πιο μακρόπνο με βάση την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως ευχαριστώ την υπατερμοστία του ΟΗΕ για την ε, εποπτεία που εξασφαλίζει ε, σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα προσφύγων. Ο κύριος Καχέμ, που είναι και αυτός μέλος της ε, αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προηγουμένω ευχαρίστησα τον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες του Οργανισμού Εθνών και εμείς ε, ετοιμάζουμε τις κοινωνίες μας ε, για να υποδεχθούν καλύτερα τους πρόσφυγες, γιατί το θέμα το προσφυγικό δεν είναι συγκυριακό, αλλά διαρθρωτικό, οπότε θα πρέπει να το φέρουμε στο επίκεντρο της προσοχής και να εξασφαλίσουμε και τους απαραίτητους πόρους. Ε, ρωτήσαμε αν θα έχουμε και τοπικού φορεί στο φόρουμ αυτό. Γιατί για να έχουμε μια κοινωνία χωρί αποκλεισμού χρειάζονται εθνικέ αποφάσει, αλλά οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ θα είναι αυτές που θα εφαρμόζουν τις αποφάσεις ε, καθημερινά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που θα έρχονται. Οπότε και ε, ως Δημαρχός του Καλέ περιμένω ε, την απάντηση της υπερσαρμοστίας που είναι καθησυχαστική ως προς τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών φορέων. Ευχαριστώ κάποιους από τους συντονιστές. Ίσως θα ήθελε το λόγο. Σίπελ, Ιντφελτ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σάντσες Αμόρ. Εγώ είμαι ο εισηγητής για την Τουρκία, οπότε περίμενα λίγο πριν να ζητήσω το λόγο. Ε, το θέμα αυτό δεν είναι ε, άμεσα συνδεδεμένο με αυτά που μας είπε ο κύριος Αντρές, αλλά θα ήθελα να θέσω το ζήτημα της Τουρκίας, που είναι μια χώρα που για πολλά χρόνια υποδέχθηκε τεράστιο αριθμό προσφύγων. Βέβαια, πολλές πτυχές πολιτικής της Τουρκίας ε, επικρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχίζονται να επικρίνονται, όπως είναι η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. Επίσης, υπάρχει και μια λανθάνωσα ανησυχία για το γεγονός ότι ίσως δίνουμε την εντύπωση ότι οι θέσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών ε, απάδουν σε ό,τι αφορά την πιθανή επιστροφή των σύρων προσφύγων από την Τουρκία. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικώ τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ήταν πολύ επικριτικά με τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας και τη, τα δημογραφικά τεχνάσματα που κάνει η Τουρκία και τη σύγκληση μιας διάσκεψης ε, δωρητών. Επίσης, ο Αρτογάν προσφέρθηκε ε, να βοηθήσει το, τους οργανισμούς του ΟΗΕ, ασκώντας όμως μία εποπτεία στην διαδικασία αυτής της επιστροφής. Γιατί υπάρχουν πολλές αμφιβολίες αν όσοι ε, επιστρέφουν στην, στην Συρία από την Τουρκία το κάνουν εκεί ο θελός. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες γι' αυτό. Ε, Επίσης, ε, ποια θα είναι η συμμετοχή της ΥΠΑ της Αρμοστίας για την εποπτεία αυτής της επιχείρησης ε, μεταφοράς ή επιστροφής. Και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη είχαν παρόμοιες θέσεις τα τελευταία χρόνια και απέτησαν το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Πώς μπορούν οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ερδογάν. Ευχαριστώ. Όσοι θέλουν να ε, ε, υποβάλουν σχόλια ή να γίνουν κάποιες ανησυχίες, θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Αλλά θα δώσω το λόγο στην κυρία Στρίκ που Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την τη ερμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το οργανωτικό της έργο και την υποστήριξη που προσφέρει στους πρόσφυγες γενικώ και θα ήθελα να ευχηθώ στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλή επιτυχία στη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους πρόσφυγες. Έχω δύο ερωτήσεις προς την Αρμοστή για τους πρόσφυγες. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζεται κυρίως στην εξωτερική ανάθεση των ευθυνών για τους ε, πρόσφυγες σε τρίτες χώρες. Μετακυλίουμε δηλαδή την ευθύνη μας προς τρίτες χώρες και βλέπετε τι αντίκτυπο έχει αυτή η μετατόπιση ευθύνης και οι τρίτες χώρες, ε, πολλές φορές που είναι χώρες διέλευσης, αντιγράφουν τη συμπεριφορά μας προς, προκειμένου να αποποιηθούν των ευθυνών τους, μεταθέτοντας την ευθύνη σε άλλους. Το, σύμφωνο, το Παγκόσμιο Σύμφωνο δίνει την ευκαιρία για, μια πιο ακριβο, ε, για πιο επιμερισμό της ευθύνη για τους πρόσφυγες. Πώς βλέπετε λοιπόν ε, τις εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ αυτής της τάσης και των επιπτώσεών της και Τη υλοποίηση του πιο μακροπρόθεσμου στόχου που είναι για δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών. Επίσης η πολιτική αυτή επισύρει επικρίσει είτε στα Ηνωμένα Έθνη είτε σε άλλα επίπεδα. Επίσης πολύ εύστοχα επισημάνατε ότι το 85% των προσφύγων είναι από ανεπτυσσόμενε χώρες και δεν ε, λαμβάνουν όλη την υποστήριξη που χρειάζονται στι περιοχέ αυτέ, λόγω των πενιχρών μέσων που έχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες για να τους περιθάλψουν. Φυσικά χρειάζεται χρηματοοικονομική υποστήριξη, αλλά σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση, δεν θα ήταν πιο σωστό να επικεντρωθούμε στους πιο ευάλωτους πρόσφυγες που χρήζουν περισσότερες βοήθειες από ό,τι μπορούν να λάβουν στην περιοχή και να επικεντρωθούν σε αυτό περισσότερο οι, οι χώρες του δυτικού κόσμου. Μήπως θα πρέπει περίπου σε αυτό το τμήμα των προσφύγων να επικεντρωθούμε στους πιο ευάλωτους δηλαδή πρόσφυγες. Ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πολύ σαφή σας παρουσίαση για το πώς έχει κατάσταση. Θέλω να κάνω δύο γρήγορες ερωτήσεις. Σωστά είπατε ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να μπουν στην κοινωνία και αυτό δεν συμβαίνει σε πολλέ περιπτώσει. Μένουν ξεχωριστά ε, επί πολλά έτη. Και αυτό αφορά κυρίως τα παιδιά που δεν έχουν καν πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό, γιατί πώς θα μπορεί να αναπληρώσει κανείς 5-6 χρόνια χαμένα από το σχολείο. Γι' αυτό λοιπόν έχουν να το εξή. Υπάρχουν κράτη-μέλη, κράτη, χώρες ε, που κάνουν ή ξεκινούν να κάνουν αυτά που θέλετε να συμβαίνουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες ε, προς τους πρόσφυγες. Πείτε μας ποια είναι η καλύτερη ή η χειρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχετε όρεξη, εν πάση περιπτώσει. Δεύτερη ερώτηση. Σε σχέση με τα άλλα μέρη του ΟΗΕ. Έχουμε χώρες που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, γιατί όπως σωστά επισημάνατε, αν υπήρχε πιο σωστή κατανομή των, του άχθους, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και τέλος, τι ε, διάκριση. Πώς ξεχωρίζετε τους πρόσφυγες από του οικονομικούς μετανάστες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σα από αυτού. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Μπίλτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα παρευρέθω στο φόρουμ για τους πρόσφυγες στη Γενέβη, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις και δεν μου έδωσαν θέση, εν περιπτώσει. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη προ του πρόσφυγες, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση που δημοσιεύτηκε πριν από κάποιες ημέρε από, τον, ε, από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του και μιλάει για 60.000 ανηλίκους πρόσφυγες ε, που έχουν ήδη ενηλικιωθεί από τότε που κατέφτασαν στην Ιταλία. 83% έφτασαν μεταξύ των 16 και 17 ετών. Είναι μια ηλικία πολύ κοντά στην ηλικία σου και αυτό δεν είναι τυχαίο προφανώ. Ε, θα ήθελα να, πω, ρωτήσω πού βασίζονται αυτέ οι εκτιμήσει. Πρόκειται για αυτά που έχουν δηλώσει οι πρόσφυγε και αυτό φυσικά μπορεί να είναι σχετικό. Μία ΜΚΟ τον προηγούμενο Ιανουάριο είπε ότι ένα τρόπο υπάρχει μόνο να διαπιστώσουμε αν είναι ανήλικοι. Να του δώσουμε, να τους κάνουμε την ερώτηση, να του ρωτήσουμε και ότι απαντήσουν. Και έχουμε νέους οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι 17 έως 19 χρονών και πάντα ε, τίθεται το θέμα αυτό για την προστασία τους και αυτό το τεστ που διαπιστώνει ακριβώς την ηλικία του παίρνει τρεις μήνες. Επίσης, σε πώς ε, δικαιολογείται τα επιπρόσθετα μέτρα υπέρ των ε, νέων αυτών ε, προσφύγων δεδομένων και των δραματικών ε, συνθήκων στις οποίες διαμένουν, για παράδειγμα, στην, στη Σικελία όπου 55% του πληθυσμού έτσι κι αλλιώς είναι ε, σε κίνδυνο φτώχειας. Και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή και στην Αιθιοπία, όπου επισκεφτήκαμε έναν καταβλισμό προσφύγων. χιλιάδες ε, άνθρωποι, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο όλες οι ερωτήσεις που ετέθησαν προς όλες τις οργανώσεις και τις ενώσεις που μας υποδέχθηκαν. Δεν ήξερε κανείς τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί εδώ και τέσσερα χρόνια και αυτό που μας είπαν ότι αυτό που θέλουμε είναι μια δουλειά, ένα σπίτι, να δουλέψουμε. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία ιδέα, καμία πρόταση για το τι θα γίνει τις, ε, τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντυπού. Σας ευχαριστώ και εγώ από πλευρά μου για την παρουσίαση και για την επισκόπηση που μας δώσατε για το πώς έχει η κατάσταση και νομίζω ότι όλα κατατεκνύουν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό να μπορέσουν να έρθουν και να συσκεφτούν όλοι αυτοί οι παράγοντες για το θέμα των προσφύγων. Ένα θέμα το οποίο αναφέρεται και όσον από τους στόχους των, της διάσκεψης. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα αναλάβουν πιο πολλά κράτη το μερίδιο της ευθύνη τους ε, για να απαλληλθεί λίγο το άχθος που βαρύνει τα υπόλοιπα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρένα. Σας ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Νάτσο για την πολιτική της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Είπατε ότι η Τουρκία αποτελεί ένα μέλος του φόρουμ. Προβλέπετε κάποια χρονική στιγμή να ζητηθεί τοποθέτηση της Τουρκίας, γιατί δεν είναι δυνατόν να, να δρά κανεί ως χώρα υποδοχής και από την άλλη και να δρά ως ε, παράγοντας αποσταθεροποίησης στη Συρία. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να το θέσουμε αυτό το ερώτημα στην Τουρκία. Το ίδιο ευχή και για την Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω κατά πόσον θα συμμετέχει στις συζητήσει. Αλλά η τραγική κατάσταση που ζούμε στην Ιεμένη με τεράστια, τεράστια όγκο εκτοπιστέντων, εσωτερικά εκτοπιστέντων και η εσωτερική κατάσταση στη χώρα, γιατί η Ιεμένη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Με βασικό παράγοντα, την Σαουδική Αραβία. Είναι παράλληλα η μεγάλη χώρα δουρήτρια ανθρωπιστική βοήθεια. Τέτοια λοιπόν ερωτήματα ανακύπτουν. Αναφερθήκατε στι βασικές αιτίε τη μετανάστευση, που συχνά ε, είναι η αποσταθεραϊοποίηση. Αυτό θα είναι θεωρητικό, μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να το θέσουμε στι χώρε αυτέ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε συχνά να τύφεται το θέμα της αιρεσιμότητας της παροχής βοήθειας. για να μπορέσουν οι χώρες ή να περιορίσουν τον πληθυσμό ή να ζητήσουν καταναστικές επιστροφές. Σήμερα, λοιπόν, στα πλαίσια της υπατησαρμοστίας έχει τεθεί το θέμα αυτό. Είπατε επίσης ότι θα είναι ενδιαφέρον να βοηθήσουμε τις χώρες προέλευσης. Μήπως θα μπορούσαμε να παρέχουμε κίνητρα, επιπρόσθετα μέτρα προς τις χώρες αυτές και όχι να μιλάμε για πραγματική ερωσιμότητα της παροχής βοήθειας στις χώρες προέλευσης. Και τέλος, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφος για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού και στις χώρες υποδοχής αλλά και στις χώρες ε, διέλευσης. Γιατί όπως είπατε οι πιο πολλοί ε, εκτοπιστέντες είναι στο ιστορικό μιας υπήρου της Αφρικής για παράδειγμα. Μάλιστα. Πολλές ερωτήσεις. Έχουμε κανέναν άλλον που θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Κάμκο. Um, Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Το... Παγκόσμιο Φόρουμ για τους πρόσφυγες προσπαθεί να πετύχει ένα καλύτερο μέλλον για τους πρόσφυγες. Ποια δόμενα έχετε για μελλοντικά σημεία πίεσης ε, ανά τον κόσμο, όπως πολιτική αστάθεια, αλλά και οι περιβαλλοντικοί παραγόντες. Όπως ε, αναφέρθηκε, στα τελευταία χρόνια η Ευρώπη ήταν απροετοίμαστη και φοβάμαι ότι ακόμα είναι. Ακόμα και αν έχουμε κάνει το σύστημα ισχυρότερο, πρέπει να ενδύνουμε τις προσπάθειες μας. Τι δεδομένα έχετε και τι τάσεις βλέπετε στα ευρήματά σας για το πώς μπορεί να βελτιώσει η Ευρώπη το σύστημά της ε, έτσι ώστε να είναι σε καλύτερη κατάσταση σε 5 ή 10 χρόνια από σήμερα. Και τι πρέπει να γίνει για την παγκόσμια συνεργασία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτά. Νομίζω. Ας ε, ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Έντρες ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τις πολλές ε, παρεμβάσεις ε, και παρεμβάσεις στήριξης, κάτι το οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερος και αντικατοπτρίζει το πνεύμα του ευαγούς αυτού Ιδρύματος. Λοιπόν, θα έλεγα πως σε σχέση με τα που είπε η κυρία Πιέρη Κέιτρη, πως ε, απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική. Εμεί έχουμε μια στρατηγική επαναγκατάσταση ε, τριών ετών και αυτό θα είναι ένα στοιχείο του φόρουμ επίσης και είναι νομίζω μια αρχή μιας ε, μακροπρόθεσμης κατάσταση. και οπωσδήποτε τελικά το απόλυτο εργαλείο προστασίας σε 85% των περιπτώσεων είναι η επαναγκατάσταση. Πάντα θα υπάρχουν κάποιε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου ή θύματα βασανιστήριων που πρέπει να πάνε σε μια τρίτη χώρα. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι αυτό το οποίο είπε η κυρία Καρέμπος. ο κύριος Καρέμπος, οι Δήμοι συχνά φέρνουν το βάρος της εισρωής προσφύγων και κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι η κατάσταση ε, κανονική και ήδη πριν από ένα έτος είχαμε μια σχετική συνάντηση και είχαμε και τις τοπικές αρχές στο φόρουμ. Όσον αφορά τον ρόλο της ε, Τουρκίας, ακούστηκαν κάποιες παρεμβάσεις. Πρέπει να αντιληφθείτε το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο του εκτοπισμού αυτό είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει κυρίως. Και πρέπει να διαχωρίσουμε στο μέτρο του δυνατού ε, την πολιτική από την ανθρωπιστική δράση, αναγνωρίζοντας πλήρως ε, το ότι απαιτείται η πολιτική δράση για να έχουμε αποτελέσματα, οπότε πλήρης διαχωρισμός δεν είναι δυνατός. Επίσης πρέπει, όπως αναγνώρισε η πρώτη παρέμβαση για την Τουρκία, να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τουρκία φιλοξενεί 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους από τη Συρία μόνο. Η επόμενη μεγαλύτερη χώρα που φιλοξενεί πρόσφυγες είναι το Πακιστάν με 1,5 εκατομμύριο. Είναι μια εξαιρετική προσέγγιση αυτή της ε, Τουρκίας και όσον αφορά τη συμπερίληψη. Το ότι επιτρέπει την ίδρυση επιχειρήσεων, 10.000 τέτοιες επιχειρήσεις που ανθούν. Πολύ θετική περίπτωση λοιπόν. Όσον αφορά δε τα πρόσφατα γεγονότα στην Βόρεια Συρία. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και ε, αυτά, θα μείνω σε αυτά για την ώρα. Το θέμα της ανάθεσης ε, σε κάποιον άλλον τώρα στις ε, φτωχότερες χώρες αν θέλετε ή να μην τους επιτρέψουμε να έρθουν στην Ευρώπη. Ε, το θέμα είναι πού βρίσκεται η ισορροπία. Και ζητάμε από όλα τα κράτη-μέλη ε, να εμπλακούν περισσότερο και αυτό περιλαμβάνει και την Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις του κόσμου με την απομόνωση. Δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία και στην βοήθεια προς τις χώρες που πάντα θα επομίζονται το μεγαλύτερο στο προσφύγων και τη ε, ε δυνατότητας να προστατευτούν οι πιο ευάλωτοι εντός της Ευρώπης. Ε, για το θέμα, ε, για την ερώτηση του κυρίου Κέλλη, σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα κατάλογο ευρωπαϊκών κρατών αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες γνωστές χώρες, δείτε ποιες έχουν πάρει τους περισσότερους πρόσφυγες ε, Ποιε δίνουν τα περισσότερα ποσά και μετά δείτε αυτές με λιγότερους πρόσφυγε και λιγότερη χρηματοδότηση. Ε, είναι μεγάλη η διαφορά μεταξύ χωρών με παρόμοιε δυνατότητε. αλλά να πω και το εξή. σε σχέση με το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Η Αιθιοπία, παραδείγματο χάρη, και έρχομαι στην επόμενη παρέμβαση, είχε μια πολιτική του να κρατά τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα ε, μακριά από τις τοπικές κοινότητες και να βασίζεται σε ανθρωπιστική βοήθεια για δεκαετίες. Τα στρατόπεδα αυτά προφανώς δεν είναι ιδεώδη. Τώρα η Αιθιοπία τον Ιανουάριο πέρασε ένα νόμο για να αντιστρέψει τελείως την πολιτική, να, επιστρέψει, να επιτρέψει πρόσφαγη στα, στους ε, πρόσβαση στα σχολεία και μιλάμε για 900.000 ανθρώπους. Αυτό απαιτεί τεράστια στήριξη από όλους τους ενδιαφερόμενους. Ανθρωπιστική ανάπτυξη, ιδιωτικό τομέα κτλ. Και αυτό ακριβώς ε, ο κόσμος θέλει να δουλέψει, το είπατε. 30.000 θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε βιομηχανικές ζώνες για πρόσφυγες στην Αιθιοπία, οπότε υπάρχει κάποια πρόοδος. Ναι, το ερώτημα του πώς ε, θα εμπλακούν περισσότερα κρατημέλη. Σας είπα, άμα τα κάνετε εντός Ευρώπης θα τα δείτε. Ποιος μπορεί να κάνει περισσότερα και παγκοσμίω βεβαίω. Υπάρχουν κάποια πλούσια κρατημέλη που δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα. Αλλά έχουμε αρκετά κράτη-μέλη ε, και έχουμε επαφές προς όλους τους δυνητικούς εταίρους που θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερη βοήθεια. Και τέλος, αντιλαμβάνομαι πλήρως ε, ακριβώς ε, το ότι κράτη-μέλη προκαλούν τον εκτοπισμό και ανησυχούν για την ανθρωπιστική πτυχή. Το αντιλαμβάνω πλήρω. Πρέπει να αντιληφθείτε κι εσεί πω και εμεί πρέπει να δουλέψουμε σε πολύ πολλωμένε καταστάσει. Ακριβώ για να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς τώρα για τα δεδομένα για μελλοντικά σημεία πίεσης Υπάρχει τεράστια συγκέντρωση αυτή τη στιγμή στο Σαχέλ. Το περιβάλλον, ε, ανασφάλεια και οι οικονομικές ε, ανισότητες ε, νομίζω τώρα δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένους αριθμούς προφανώς κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να υπάρχει ένας προγραμματισμός και με το Συμβουλίο της Ασφαλείας. Αυτό θα ήθελα να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν επανέλθω στο βήμα, ε, υπάρχει νομίζω τώρα λίγος χρόνος για να μας πει η Κομισιόν την άποψη της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τους πρόσφυγες. Ε, θέλει ο εκπρόσωπος ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να μιλήσει. Η Κομισιόν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνική, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Θα ήθελα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την ύπατη αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για του Πρόσφυγε για το, την επικέντρωση του, του φόρουμ στους εκτοπιστέντες και στους πρόσφυγες Έχουμε ιδιαίτερη εταιρική σχέση, ιδιαίτερα για τον αναγκαστικό εκτοπισμό με την υπατιαρμοστία. Θεωρούμε ότι αυτό το Παγκόσμιο Φόρουμ για τους πρόσφυγες θα είναι μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια δυναμική και να θετήσουμε πιο εύκολα τους, να υλοποιήσουμε πιο εύκολα τους στόχους του Παγκόσμιου Συμφώνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των προσφύγων. Επίσης, με το φόρουμ θα συνειδητοποιήσουμε τα επιτεύγματα και θα προβούμε σε μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, θα συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση μεμονωμένων χωρών, συγκεκριμένων περιφερειών και παγκοσμίω. Επίσης, θα βοηθήσουμε την ε, διεθνή κοινότητα να αναζητήσει λύσεις για να αλαφρύνουμε ε, ε, τα πάνδυνα που υφίστανται οι πρόσφυγες. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό δωρητή παγκοσμίω, αλλά και βασικός παράγοντα στην προστασία των προσφύγων, την παροχή αρρωγή στους πρόσφυγε και την προσφορά λύσεων. Και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την ηγετική μα θέση και να την αναδείξουμε και στο Παγκόσμιο Φόρουμ. Ε, συνεχίζονται οι προετοιμασίε μα ε, εν ώψη του Φόρουμ και μάλιστα ε, τέσσερις από τις έξι τομείς θα τους ε, χρηματοδοτήσουμε και εμείς και θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε τις πολιτικές μας ό,τι αφορά την παιδεία, την προστασία σε περίπτωση κρίσης, στους ε, αναγκαστικούς εκτοπισμούς και θέλουμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες ε, υιοθετώντα την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Προσβλέπουμε σε αυτή τη συμμετοχή μα στο Παγκόσμιο Φόρουμ για του Πρόσφυγε και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μα με την Υπετερμοστή για του Πρόσφυγε και πέραν του φόρουμ αυτού, προκειμένου να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το σύστημα της του αναγκαστικού εκτοπισμού, που όπως είπατε είναι ένα διεθνές πρόβλημα που χρήζει ε, ανάληψη συλλογικής ευθύνης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στη συνεργασία με την υπατερμοστία και μετά το φόρουμ να προσπαθούμε να διαθετήσουμε το ζήτημα του αναγκαστικού εκτοπισμού. Από το πάνελ μας θέλει κανείς το λόγο για να αντλήσει κάποια συμπεράσματα από τη συζήτηση ο Τωμά Τομπέ από την Επιτροπή Ανάπτυξη. Ευχαριστώ την Υπατιαρμοστή για την ανταλλαγή απόψεων. Σίγουρα το ζήτημα είναι πολύ σύνθετο και εξαιρετικά δύσκολο, αλλά είναι σημαντικό στο μέλλον να έχουμε κάποια πρόοδο. Σωστά είπε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ότι θα πρέπει στα αναπτυξιακά μα σχέδια να συμπεριλάβουμε και τους ε, πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλο που έχουμε διάσταση απόψεων ακόμη και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μερικά ζητήματα, νομίζω ότι συμφωνούμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει αυτό τον ηγετικό της ρόλο ε, στην προστασία και υπεράσπιση της πολυμέρειας. Θα ήθελα να ευχηθώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καλή τυχή και αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι τα έργα και όχι τα λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. με ιδιαίτερο τη συμμετοχή σας και θα ήθελα να μεριμνήσουμε ώστε αυτό το φόρουμ της Γενέβης ε, που θα προσπαθήσει να υλοποιήσει το παγκόσμιο σύμφωνα για τους πρόσφυγες ε, θα είναι ευκαιρία για να κάνουμε τη διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και της παραπληροφόρησης. Ε, γιατί μερικές φορές η συζήτηση έχει ε, δηλητηριαστεί από τοξικά και πλαστά, τοξικές και πλαστές ειδήσει. Εδώ μιλούμε για... θα πρέπει να δούμε ποιοι, ποιοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί των μετακινήσεων αυτών. Έχουμε το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθροδιακινητών. Θα πρέπει να το α, καταρρύψουμε και έχει, έχουν κυκλοφορήσει τέτοιες α, ανεδαφικές φήμες για την αποκαλούμενη προσφυγική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συχνά έχει προβληθεί και παρουσιαστεί ως απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα τέτοιο δεν ισχύει. Όλα αυτά είναι αβάσιμα, είναι παραπληροφόρηση και μια τέτοια εξτρατεία δεν συνάδει με τις ε, αρχέ και τις αξίε Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταστρατηγεί το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Γι' αυτό και χαίρομαι που έχουμε τέτοιε ευκαιρίε να ανταλλάσσουμε απόψει για τις βέλτιστες πρακτικέ, προκειμένου να βελτιώσουμε, όχι μόνο να ενισχύσουμε, αλλά να βελτιώσουμε την ποιότητα τη ε, Ευρωπαϊκή απόκριση σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που δεν πρόκειται να περατωθεί στο εγγύς μέλλον ή να διακοπεί. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόσο προσιλωμένο και θέλει να είναι ενεργός παράγοντας, όχι απλώς μάρτυρας, αλλά σημαντικός παράγοντας στις συζητήσεις και στα έργα που θα ακολουθήσουν. Συνεχίζουμε αμέσως μετά την το ξεπροβόδισμα των καλεσμένων μας με την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών. Σας ευχαριστώ. If you will. Χωρίς άλλη καθυστέρηση. Συνεχίζουμε ακάθεκτη στο επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης, το υπαριθμό 14, με θέμα την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας του 2013. Παρακαλώ ησυχία. Βοήθεια, ησυχία παρακαλώ. βοήθειά μας θα μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε, με τη βοήθειά σας θα μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε την ημερήσια διάταξη. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο σημείο 14, έκθεση Επιτροπής για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο στα πλαίσια ποινική διαδικασία και διαδικασία εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη, καθώ και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωση τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρηση τη ελευθερία του και με το δικαίωμα επικοινωνία με τρίτα πρόσωπα και με προξενικέ αρχέ κατά τη διάρκεια τη στέρηση τη ελευθερία. Εδώ μιλούμε για την εφαρμογή της οδηγίας του 2013 και ήταν ένα από τα μέτρα που, που υιοθετήθηκαν μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Οδικού Χάρτη του Συμβουλίου του 2009 για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων. Είχαμε το πακέτο, τη δέσμη μέτρων των δικονομικών δικαιωμάτων και στα πλαίσια του πακέτου αυτού έχουμε υιοθετήσει έξι οδηγίες που προσπαθούν να υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική και να ενισχύσουν τα δικονομικά δικαιώματα με νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Ενωσιακού Δικαίου. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στα πλαίσια αυτής της δέσμης μέτρων για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων. Είχαμε και την τρίτη οδηγία που εγκρίθηκε για τα δικαιώματα μετάφραση και διερμηνίας σε ποινικέ δίκες και δικαίωμα σε ενημέρωση για, ποινικής, για την ποινική δικονομία. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ακόμη υψηλότερε προδιαγραφέ, το δικαίωμα σε δικηγόρο, ω αναφέρετο και απόλυτο δικαίωμα σε όλα τα κοινοτικά κράτη-μέλη. Μετά μας την επιμόνη του Συμβουλίου για τις εξαιρέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 5 και 6 ε, με βάση γεωγραφικά προβλήματα και περιορισμένες εξαιρέσεις σε προκατακτική αστυνομική φάση, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς εφαρμόστηκαν αυτές οι εξαιρέσεις στο εθνικό δίκαιο και σε πόσες χώρες μέλη εφαρμόστηκαν. Θα ακούσουμε λοιπόν ε, την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Παρακαλώ, το λόγο έχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλησπέρα σα και σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την ε, αξιολόγησή μας ε, για την εφαρμογή της οδηγίας για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Και δεν ε, αναφέρεται μόνο στην πρόσβαση στο δικηγόρο οδηγία, αλλά και στο σημαντικό θέμα της επικοινωνίας, σε περίπτωση που κάποιος έχει στερηθεί ε, της ελευθερίας του. Έχουμε μάλιστα υποβάλει τη σχετική έκθεση ε, εμπρόθεσμα και λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Η προθεσμία λήγει τέλη Νοεμβρίου. Εμείς εκπονήσαμε ε, την έκθεση ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου και ακριβώς την ίδια μέρα ο Οργανισμός ε, Θεμελιδών Δικαιωμάτων της Βιέννης υπέβαλε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με το ίδιο αντικείμενο. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε που μας υπενθυμίσατε ε, το γενικό πλαίσιο του νομοθετικού προγράμματος ε, και της μέρος, μέρος το οποίο είναι και η οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο και μάλιστα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα και θα ε, θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό το νομοθετικό σχέδιο εστέφθη με μεγάλη επιτυχία. Και αν συγκρίνουμε την κατάσταση με τις έξι οδηγίες που υιοθετήθηκαν μετά τον οδικό χάρτη του Συμβουλίου του 2009 που μας αναφέρατε, βλέπουμε ότι έχουμε πια πολύ υψηλότερα πρότυπα και προδιαγραφές σε σχέση με αυτά που είχε προτείνει νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004 δηλαδή με τη θέση πλαίσιο για τα δικονομικά δικαιώματα. Η απόφαση πλαίσιο που συζητήθηκε τότε στο Συμβούλιο χωρίς συμμετοχή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, είχε γίνει τότε γιατί τότε δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και τελικά η πρόταση τότε είχε κολλήσει στο Συμβούλιο λόγω της ανάγκης της ε, ομοφωνίας για την υιοθέτηση της απόφασης. Και αυτό είναι σημαντικό υπόβαθρο να το έχουμε υπόψη. Ε, σημαντικό ιστορικό. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την οδηγία, κάποια κρατημέλη ε, εφάρμοσαν την οδηγία αυτή για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο λόγω της νομολογίας επί της υπόθεσης Σαλντούς. Και πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η νομολογία, η απόφαση της υπόθεσης Αλντούς. Γιατί το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε αυτή τη σημαντική απόφαση εξηγώντας ότι η νομική εκπροσώπηση από δικηγόρο θα πρέπει να είναι δυνατή από την πρώτη ανάκριση, σε πολύ πρώιμες φάσεις δηλαδή της αστυνομικής έρευνας και ανάκρισης. Επίσης, ε, η απόφαση αυτή υπογραμμίζει αν δεν εξασφαλιστεί τέτοια πρόσβαση σε δικηγόρο από τα πρώιμα στάδια, θα έχει παραβιαστεί το δικαίωμα σε υπεράσπιση και μάλιστα ανεπανόρθωτα. Και μάλιστα αυτό συνέβη πριν τις ε, ε, διαδικασίες για την οδηγία και ακολούθησε η εφαρμογή τέτοιων ε, νομοθετικής διάταξη από πολλά κράτη-μέλη. Στη συνέχεια, υιοθετήσαμε το 2013 την οδηγία για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, πολύ νωρίτερα από την δίδυμη οδηγία για την ε, νομική αρρωγή, που ακολούθησε το 2019. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χωρίσει αυτά τα μέτρα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δικηγόρο και σε νομική δικαστική αρρωγή, λόγω της οικονομικής κρίσης που σοβούσε τότε και λόγω της περιπλοκότητας του ζητήματος. Οπότε συνεχίσαμε την προσέγγιση μας βάσει το δίκου χάρτη και υιοθετήσαμε μια κλιμακωτή σταδιακή προσέγγιση και τελικά υιοθετήσαμε αυτές τις έξι οδηγίες. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο, η περίοδος μεταφοράς ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και έκτοτε αρχίσαμε την αξιολόγησή μας, τον έλεγχο μας. Ήδη στην περίοδο εφαρμογής βοηθήσαμε τα κρατημέλη οργανώνοντας συναντήσεις με εμπειρογνώμονες και εκεί παρουσιάσαμε την οδηγία και πολλά σχέδια και προγράμματα που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει την, τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή. Αυτό άλλωστε συνέβη και με τις έξι οδηγίες του πακέτου. Μετά την α, παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκκίνησε εννέα διαδικασίες επί για μη κοινοποίηση των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας. Γιατί εννέα χώρες δεν υπέβαλαν ε, ανακοίνωση για εφαρμοστικά μέτρα μετά την πάροδο της προθεσμίας. Και μάλιστα τρεις από τις εννέα διαδικασίες που εκκρεμούν ακόμη. Και τώρα μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησαμε, ε, εκπονήσαμε τη μελέτη περί εφαρμογής, την έκθεση αυτή που σας παρουσιάζω σήμερα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα διάφορα άρθρα της οδηγίας και στο πλαίσιο των διαφορών διατάξεων να σταθώ σε κάποια θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ξεκινάμε εδώ με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα ε, πρόσβαση δικηγόρο στο πλαίσιο ποινική διαδικασία. Άρθρο 2. Το σημείο αφετηρίας για την γέννηση των δικαιωμάτων είναι η επίσημη κοινοποίηση ή με άλλο τρόπο κοινοποίηση της έναρξης των ποινικών διαδικασιών κατά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και μάλιστα εσκεμένα οι συνομοθέτες επέλεξαν αυτή τη χρονική στιγμή χωρίς να αναφέρονται στην επίσημη πράξη κατηγορίας, στην απαγγελία της κατηγορίας. Αυτό θα πρέπει να προέλθει από πρόσωπο των αρχών επιβολής του νόμου. Γενικώ αυτή η διαδικασία ε, και το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σωστά είτε από νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται σε τέτοιες δραστηριότητες είτε από διατάξεις που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και που εξασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα ήδη σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας. Βέβαια, ε, μας προβληματίζει η κατάσταση σε δύο-τρεις χώρες που εξακολουθούν να αναφέρονται σε επίσημη απαγγελία κατηγορίας. Και εδώ υπάρχουν αφιβολίες για το κατά πόσο οι κανόνες αυτοί ισχύουν από τη στιγμή στέρηση της ελευθερίας και αφήνουν ανοιχτό το θέμα το κατά πόσο η πρόσβαση σε δικηγόρο ε, ισχύει ακόμη και όταν κάποιος δεν έχει στερηθεί της ελευθερίας του. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, άρθρο 2.2, αυτό προβλέπει ότι ισχύει από τη στιγμή της σύλληψης. Τα περισσότερα κράτη-μέλη πρότειναν μια εφαρμογή κατά αναλογία, μουτά της μουτάντης, ώστε να προσαρμοστούν στις διαδικασίες ε, του Ευρωπαϊκού Ενδάλματος Σύλληψης και με βάση ε, την ποινική δικονομία. Μερικές φορές ίσως δεν καλύπτονται όλα τα δικαιώματα. Επόμενη διαφάνεια. Πάμε στο βασικό δικαίωμα της πρόσβασης σε δικηγόρο, άρθρο 3 της οδηγίας. Το άρθρο 3 προβλέπει το σημείο αφετηρίας και το περιεχόμενο του δικαιώματος. Επίσης, ε, τονίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το άρθρο και προκύπτει από την ομολογία Σαλντούς ότι θα πρέπει να δίνεται αυτό το δικαίωμα και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και ιδιαίτερα όταν κάποιος στερείται της ελευθερίας του. Τώρα, δεν είναι σαφές αν θα πρέπει να ισχύει και πριν την ανάκριση από τις αρχές. Και στην περίπτωση αυτή είχαμε αμφιβολίες για το κατά πόσο το δικαίωμα θα πρέπει να ισχύει και πριν ε, την ανάκριση, ώστε να ετοιμαστεί με το δικηγόρο του ο ύποπτος εν ε, της έρευνας από τις αρχές. Επίσης, ε, δεν θα, πρόκειται, ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την στέρηση της ελευθερίας. Αυτό το άρθρο το εφαρμόζουν χωρίς πρόβλημα τα περισσότερα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συμβουλή δικηγόρου πριν την σύλληψη, Ε, και πώς διαρκεί αυτή η συνομιλία με τον δικηγόρο. Συνήθως είναι μισή ώρα. Έχουν κάποιες χώρες, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο διεξοδικά. Πάντως, όπως είπε και προηγουμένως, θα πρέπει να μιλούμε για τα θέματα της εξαίρεσης από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο. Αυτό το θυμάμαι γιατί ήμουν στην διαπραγματευτική ομάδα τότε ε, ήταν ένα σημείο που συζητήθηκε εκτενέστατα μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, εντό των δύο οργάνων, ξεχωριστά δηλαδή και μεταξύ του. Και θυμάμαι ότι ήταν ε, ένα από τα πιο δύσκολα σημεία η εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας μεταξύ του υπόπτου ή του κατηγορουμένου και του δικηγόρου του. Και επίμαχο ζήτημα ήταν και οι εξαιρέσει. Και ήταν από τα πιο δύσκολα θέματα που μόνο στους τριμερείς, τελευταίους διαλόγους διαθετήθηκαν. Και όπως είπατε σωστά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε ιδιαίτερος σε μια διεξοδική ανάλυση του θέματος αυτού των εξαιρέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση που υποβάλλουμε. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρατών μελών που χρησιμοποίησαν αυτή τη δυνατότητα εξαίρεσης, μπορούμε να πούμε ότι 4 πέμπτα των κρατών μελών εφάρμοσαν τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγραφός 6. Επίσης το 3-6 όντως επιτρέπει κάποιες εξαιρέσεις υπό αυστηρούς όρους όμως. Σε ό,τι αφορά τη φυσική, σωματική αικαιρεότητα τη ζωή του ή κάποιες κατεπίγουσες έρευνες. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στα κράτη-μέλη, πολλές χώρες μετέφεραν σχεδόν πιστά το περιεχόμενο της οδηγίας ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις. Κατά γράμμα ή ε, με παρεφερές πολύ περιεχόμενο. Ε, και αυτός προς τις δυνατότητες, αλλά μερικές φορές τα κριτήρια ίσως είναι αμφισβητήσιμα, γιατί αναφέροντα σε κάποιους γενικούς κινδύνους παρεμπόδισης ε, των αποδεικτικών στοιχείων ή παρεμποδίζοντας την έρευνα ή την επιτυχία, την επιτυχία κατάληξη της έρευνας. Μερικές φορές μας προβληματίζει ο σύνδεσμος αυτών των απαιτήσεων με τις προϋποθέσεις της οδηγίας. Στην οδηγία μιλούσαμε για τη δικαιολόγητη παράταση του χρόνου κράτησης ή ανωτέρα βία ή σε περίπτωση που η καθυστέρηση των ερευνητικών δράσεων θεωρούνταν ότι διακύβευαν την ασφάλεια. Άλλες διατάξεις που αποτελούσαν χαρακτηριστικές εξαιρέσεις θα έπρεπε να αναλυθούν. Για παράδειγμα, κάποιες διατάξεις που προβλέπουν ότι όταν αποδεικνύεται ότι ενημερώθηκε ο, ο δικηγόρος για την ημερομηνία μιας δράσης, οι αρχές θα μπορούσαν να προχωρήσουν ή κάποιες διατάξεις που αναφέρονταν σε μία πράξη που δεν θα μπορούσε να αναβληθεί ή που δεν θα γίνονταν κατάλληλη ενημέρωση του δικαστικού πλήρου εξουσίου. Επίσης, ένα τρίτο θέμα που χρήζει ανάλυση είναι τα χρονικά περιθώρια για την ε, παρουσία του δικηγόρου. Μερικές φορές θεωρήθηκα πολύ περιοριστικά. Πάντως, στα περισσότερα κράτη-μέλη και στα, ακόμη και στα κράτη-μέλη που έχουν κάποια χρονικά περιθώρια, στο μεταξύ προβλέπεται η έγκαιρη προειδοποίηση, ειδοποίηση μάλλον του δικηγόρου, η έγκαιρη ανακοίνωση στο δικηγόρο και τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται ε, να γίνει γρήγορα η έρευνα ή η ανάκριση σε συγκεκριμένα περιθώρια, τότε ή για, να υποβληθεί, παραπευθεί στο δικαστήριο η υπόθεση, τότε υπάρχουν ειδικέ διατάξεις για τα χρονικά περιθώρια. Πάντως και το θέμα των χρονικών ορίων θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω. The other topic... Στην επόμενη διαφάνεια, το άλλο θέμα το οποίο σας παρακαλώ, λέει ο ε, παρακαλούμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταλαβαίνουμε ότι κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε, αλλά έχουμε και την επόμενη ε, παρουσίαση στις 4 και θα πρέπει να έχουμε κάποιο περιθώριο και τα μέλη να θέσουν ερωτήσεις. Θα παρουσιάσετε παρακαλώ να συνοψίσετε, να ολοκληρώνετε. Ναι, ναι, ναι. Νόμιζα ότι είχα μισή ώρα στη διάθεσή μου, αλλά προφανώς πρέπει να βιαστώ. Νόμιζα ότι είχα μισή ώρα, μισή ώρα στη διάθεσή μου οι παρουσιάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή ενώπιον του Κοινοβουλίου ουσιαστικά έχουν ω σκοπό τη διεξαγωγή συζήτηση, όχι απλά τη δήλωση ζητημάτων, σε ό,τι αφορά το απόρριτο της επικοινωνία, ε, Μια αρχή η οποία ήταν πάρα πολύ βασική και την οποία επαναλαμβάνει και κατοχυρώνει η οδηγία. Διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Ένα άλλο θέμα όπου είχαμε πιο πολλές ανησυχίες ήταν το θέμα της ε, εξαίρεσης. Θα το δούμε και στην επόμενη διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους, σε δικηγόρο στην ε, Ευρωπαϊκή Διαδικασία Σύλληψης, στο κράτος μέλος το εκτελεστικό υπήρχε συμμόρφωση με το θέμα αυτό. Ετύφεται το θέμα του κράτους μέλους έκδοσης. Εδώ ο μηχανισμός συνεργασίας σε κάποιες περιπτώσεις υστερεί. Το θέμα της επικοινωνίας ε, μετά τη σύλληψη, εδώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Μπορείτε να διαβάσετε και τις ε, διαφάνειες μετά, άμα θέλετε. Αυτή η επαφή πρέπει να είναι δυνατή κατά τη διάρκεια τη σύλληψη, χωρί οποιαδήποτε καθυστέρηση. Εδώ τίθεται και το θέμα του πεδίου ισχύω τη οδηγία. Εδώ, εδώ ενδεχομένω να έχουμε κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τι αποκλήσεις, τι εξαιρέσει που αφορούν οκτώ κρατημέλη. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, 2 και 4, πολύ σημαντικές ε, διατάξεις για κατηγορούμενους κάτω των 18. Εδώ είναι πολύ σημαντική η διάταξη αυτή. Εδώ προκαλούνται ανησυχίε. Γιατί σε κάποιε περιπτώσει ε, η διαδικασία ενημέρωση κάποιου άλλου κατάλληλου ατόμου, όταν ε, δεν υπάρχει άτομο υπεύθυνο για το παιδί, ή ενδεχομένως να λαμβάνεται υπόψη η ενδεχομένω να υπάρχει ενημέρωση του γονέα χωρίς ε, καθυστέρηση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, επαφή με τρίτα άτομα, η επαφή και με τις προξενικές αρχές και με τρίτα άτομα. Η επικοινωνία με τρίτα, κράτη, πρόσωπα υπάρχει σε όλα τα κράτη, μέλη. Σε κάποια κράτη-μέλη ενδεχομένως να προκαλείται να ξεκινά αργότερα. Ιδιαίτερα άμα πρόκειται για κράτη-μέλη που έχουν εκφράσει ανησυχίε σε ό,τι αφορά την ε, άμεση αυτή επικοινωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα την επικοινωνία με τις προξενικές αρχές, συχνά βλέπουμε άμεση ισχύ της ε, Σύμβαση της Βιέννης που σχετίζεται με το άρθρο 7 της οδηγίας. Εδώ ήταν σωστή ως επιτοπλίστων η εφαρμογή. Στην τελευταία διαφάνεια, μάλλον την πρώτη τελευταία. Τα βασικά λοιπόν θέματα τα οποία παραμένουν έκρεμοι. Αυτό ήταν και το δικό μας συμπέρασμα. Έχουν να κάνουν με το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Διτάξεις ε, αυτές που αντίφονται σε ισχύ μόνο μετά από τη σύλληψη του ατόμου, θέματα για τις ε, ε, εξαιρέσεις, θέματα για τις αποκλήσεις και το δικαίωμα πρόσβαση δικηγόρο στο κράτο μέλο έκδοση. Θα κλείσω στο σημείο αυτό και την τελευταία διαφάνεια θα δείτε τη σημασία τη οδηγία αυτή και των επόμενων ε, οδηγιών για την νομική αρρωγή και για τα παιδιά, τους ανηλικούς όλους ιδιαιτέρους και να έχουμε υπόψη ότι αυτές οι οδηγίες ε, είναι πολύ σχετικές και συνδέονται μία με την άλλη. Θα είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να εφαρμοστεί η οδηγία για την δυναμική οργή. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ και εγώ για την υπομονή σα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ναι, μα μισή ώρα ήταν η ώρα που προβλεπόταν για όλο το θέμα αυτό και για τι συζητήσει. Και έχουμε κάποιου βουλευτέ που θέλουν να πάρουν το λόγο. Τρει. Αν θέλει κανεί άλλο να κάνει κάποια ερώτηση, να μα το πει, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Δεν μπορούμε να, περιμένει, να αφήσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνη τη Λιθουανία να περιμένει. Η κυρία Σίπερ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την έκθεση και ήδη στην εισαγωγή της ε, μας έδειξε πόσα προβλήματα έχουμε ακόμα μετά από έξι χρόνια από την έγκριση αυτής της οδηγίας. Αυτό ισχύει και για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δεδομένο. Για την εμπιστευτικότητα της ε, συνεννόησης με τον δικηγόρο και επίσης για τις προθεσμίες που έχουν ε, οι δικηγόροι να ενημερώσουν ότι δεν υπάρχει δικη δίκη. Και βεβαίως συχνά κατά τη διάρκεια της σύλληψης ενθαρρύνονται οι άνθρωποι να αρνηθούν το δικαίωμά τους σε δικηγόρο ή έχουν ελάχιστες πληροφορίες. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής. ειναι η εξη έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάση, πόσες από αυτές είναι ακόμα ανοιχτές, αφορούν λίγο πολύ τα ίδια πράγματα όλες και πόσες χώρες ακόμα δεν έχουν Εφαρμόστε την οδηγία. Ευχαριστώ κύριο Σαρσαρέχο. Muy brevemente, eh, señor eh, Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα από τα εκκρεμή θέματα είναι η πρόσβαση σε δικηγόρο στα κράτη-μέλη που εκδίδουν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Μπορείτε να μας το αναπτύξετε αυτό πιο διεξοδικά, αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Κυρίε Κινίτσι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την ε, Κομισιόν. Έχω ένα ερώτημα συγκεκριμένο για τις εγγυήσεις που αφορούν τους ανήλικους που βρίσκονται στο άρθρο 5, παραγραφός 2 και 4 της οδηγίας και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν εάν έχει στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται για τους ε, ανηλίκους ε, ή άλλες ε, περιπτώσεις όπως οι γυναίκες ή έγκες οι οποίες πρέπει να ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της κράτησης και βεβαίως αν δούμε τη σελίδα 14 της έκθεσης βλέπουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη η νομοθεσία δεν προβλέπει σαφείς μηχανισμούς που θα λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον ε, του παιδιού σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ρωτήσω την Κομισιόν αν υπάρχει κάποιος αριθμός για τα κράτη-μέλη αυτά και κυρίως ε, τι σκοπεύει να κάνει για να εργοποιήσει αυτές τις διατάξεις, ειδικά σε σχέση με την οδηγία 2016 καθώς 800 που έχει ενισχύσει τις προστασίες των ανηλίκων. Ευχαριστώ. Κυρία Μπορέκ, ευχαριστώ. Το άρθρο 13 της οδηγίας λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες ανάγκες ευπαθών κατηγορουμένων. Η έκθεση της Κομισιόν λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν ειδικέ διατάξεις για ανάπηρους και παιδιά. Δεν αναφέρει άλλους λόγους για ευπαθή άτομα γνωρίζει η Κομισιόν αν υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία προηγούμενο ψυχολογικό τραύμα, παραδείγματο χάρη να από ενδοοικογενειακή βία αποτελεί λόγο για να θεωρηθεί κάποιος ευπαθής. Μάλιστα, δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει το λόγο. Οπότε παρακαλώ την Κομισιόν. Είδατε ότι οι βουλευτές ε, ήταν σύντομοι. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να απαντήσετε σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίω για εμάς είναι σημαντικό να γίνει σωστά η εφαρμογή της οδηγίας αλλά θα ήθελα να τονίσω πως συνολικά έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα εδώ πέρα να πω πως η Κομισιόν είναι θέμα των συνθήκων και γνωρίζουμε τον ρόλο μας αυτόν, οπότε όπως ε, είπε και ο κύριος Ρεντέρ, ο υποψήφιος επίτροπος, θα παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη των μέσων αυτών και της οδηγίας αυτής οπωσδήποτε. Και δεν θα διστάσουμε να ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Υπάρχει βεβαίως ε, το θέμα της πρόσβασης σε δικηγόρο στο κράτος μέλος που εκδίδει το ένταλμα, αλλά δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό περιπτώσεων όπου ο ε, μηχανισμός ε, που αφορά τα συμφέροντα του παιδιού και ενημέρωση κάποιου άλλου ενηλίκου θα εφαρμοστεί όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ε, έχουμε κάποιες ερωτήσεις ε, που αφορούν 10 κράτη-μέλη. Το άρθρο 13 για τους ευπαθείς, ε, τα ευπαθή άτομα. Εδώ πέρα θα ήθελα να πω πως έχει υπάρξει μια σύσταση της Κομισιόν για τα ευπαθή άτομα που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πως μιλάμε για μια ετερόκλητη ομάδα και είναι δύσκολο να έχουμε ακριβείς ε, διατάξεις. Ευχαριστώ, ελπίζω να ήμουν σύντομη. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ε, να μας στείλετε την παρουσίαση αυτή σε όλους τους βουλευτές για να μπορούν να αναλύσουν αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Περνάμε στο επόμενο. Άλλη μια παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Λιθουανίας, τον κύριο Ελβίνας Γιανκεβίτσιους. Σας καλωσορίζουμε. Κύριε Υπουργέ, And we're also welcoming the participation in this point in the order of the day. Ε, καλωσορίζουμε επίσης ε, τον κύριο Βάλτα Πασίλης, ο Υπουργό Δικαιοσύνη, ε, ο Γενικό Αγγελέα, με και ο Νέργιο Μέλτση, ο οποίο είναι ε, πρόεδρο ε, του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Κάουνα. Θα διαφωτίσουμε και τα μέλη της Επιτροπής μας για το ευαίσθητο αυτό ζήτημα για μία ώρα. Μία ώρα έχουμε προγραμματίσει. Παρακαλώ να το έχετε κατά νου. Οπωσδήποτε είναι χάρα μας που έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Γιανκεβίτσιους για αυτό το λεπτό θέμα. Στις 24 Ιουλίου ως πρόεδρος της Επιτροπής έλαβα μία επιστολή από τον Υπουργό που επισήμενε στο Κοινοβούλιο ολόκληρο και στην Επιτροπή μας την ε, λεγόμενη υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου που περιλαμβάνει διώξεις ε, δικαστών και εισαγγελέων από την Ρωσική Ομοσπονδία. Συναντήθηκα λοιπόν με τον κύριο Υπουργό, μου εξήγησε λεπτόμερος και ο Υπουργό προσφέρθηκε να έρθει στην Επιτροπή μας να τα εξηγήσει αυτά και ελήφθη απόφαση από τους ε, συντονιστές υπό το φως ε, της εμπλοκής ε, της Επιτροπής Εξωτερικών βεβαίως, καθώς το θέμα αφορά τις ε, σχέσεις με την Ρωσία. Ναι, έχουμε προσκαλέσει και τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών. Τι είναι λοιπόν αυτή η υπόθεση. Το 1991, στις 13 Ιανουαρίου, είχαμε ματηρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών για την εξαρτησία της ε, χώρας και σοβιετικών στρατευμάτων στο κτίριο της ε, τηλεόρασης ε, στο Βιλνίους. Μια, ένα, μια δραματική στιγμή στην ιστορία της χώρας. 14 άμαχοι σκοτώθηκαν και 702 τραυματίστηκαν. Τον Μάρτιο φέτος ε, το Περιφυρακό Δικαστήριο του Βίλνιους είπε ότι τα γεγονότα αυτά ήταν επιθετική ενέργεια της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Λιθουανίας και άρα θεώρησε ότι ο κύριος Δημήτρη Γιάτσοφ, τότε υπουργό Αμήνης Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και 60 ακόμα άτομα, αξιωματούχοι της Σοβιετικής Ένωσης, ε, ε, ήταν ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τα γεγονότα της 13ης Ιανουαρίου. Με έχουν ενημερώσει πως αναζητήθηκε η δικαστική συνεργασία με την Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά μόνο 5 από τα 289 αιτήματα ε, ικανοποιήθηκαν μερικώς. Επιπλέον, το 2018 η Εξεταστική Επιτροπή της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας ε, ξεκίνησε ποινικέ διώξεις κατά των εισαγγελίων της Λιθουανίας που ερεύνησαν την υπόθεση. Και φέτος κατηγορήθηκαν οι δικαστές αυτοί σε ποινικό δικαστήριο. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της ε, Λιθουανίας και ο Γενικός Εισαγγελέα και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Κάουνας και τους βουλευτέ βεβαίω μετά. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την εισαγωγή. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, σα είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα παρουσιάσω και να συζητήσουμε τι πρόσφατε δράσει τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά Λιθουανών δικαστών και εισαγγελέων που συμμετείχαν στις έρευνες των τραγικών γεγονότων της 13 η Ιανουαρίου του 1991 στο Βίλνιους, όταν η Σοβιετική Ένωση προσπάθησε να συντρίψει την πρόσφατα ανακτήσα ανεξαρτησία του έθνους μας. Είναι σημαντικό όμως να δούμε αυτά τα γεγονότα στο ιστορικό τους ε, πλαίσιο μετά την ολοκλήρωση ε, τη, του πρωτοκόλλου του Μολότοφ Ρίβεντροφ και των μυστικών πρωτοκόλλων ε, του, 49, του, του 49 όταν η Σοβιετική Ένωση κατέλαβε τις ανεξάρτητες δημοκρατίες της Λιθουανίας, Εστονίας και Λετωνίας μετά την Διακήρυξαν εξαρτησία στις 11 Μαρτίου ε, του 1991, η, η Σοβιετική Ένωση έκανε μια επιθετική δράση κατά της Λιθουανίας στις 13 Ιανουαρίου του 1991. Ο Σοβιετικός στρατός ε, έκανε στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, κατά του λαού της Λιθουανίας. Και μάλιστα έχω και διαφάνειες, αν μου επιτρέπετε. Τα σοβιετικά στρατεύματα αποφάσισαν να ε, κλονίσουν την ελευθερία μας, να διαταράξουν την τάξη μας. Όπως ξέρετε όμως δεν τα κατάφεραν. Παρ' όλα αυτά τότε προσπάθησαν και κατέβαλαν το, ε, το Υπουργείο Άμυνας, ε, τον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίλνιους και τον τηλεοπτικό σταθμό του Βίλνιους και προσπάθησαν τα σοβιετικά στρατεύματα να καταλάβουν και τη Λιθουανική Βουλή και μάλιστα τότε ένα μεγάλο πλήθος άμαχων, άοπλων κατέβηκαν στους δρόμους για να προστατεύσουν τους θεσμούς μας. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά όλοι από κοινού ε, στο, μέσα στον κρύο χειμώνα διαδηλώναμε ελπίζοντας ότι τίποτα θα συμβεί. Και η νύχτα αυτή ήταν η 13η Ιανουαρίου του 1991 Είχαμε όμως τραγικά γεγονότα στον τηλεοπτικό σταθμό του Βίλνιους. Είχαμε επίθεση με εκατοντάδες τραυματίες και τα στρατεύματα και τα τάγκ εμφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι. Σταμάτησαν τον κόσμο, δεν σταμάτησαν να όμως ε, τους πυροβολισμούς ε, ε, προέλασαν και κατέλαβαν και το τηλεοπτικό σταθμό. Τότε είχαμε θανάτους και εκατοντάδες τραυματίες λόγω της επιθετικής δράσης του Σοβιετικού στρατού τη νύχτα εκείνη της 13ης Ιανουαρίου που ακόμη μας πονάει. Και φέτος το Μάρτιο το Λιθουανικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σε μια ποινική υπόθεση για τα γεγονότα της 13ης Ιανουαρίου του 1991. Και μάλιστα με βάση την απόφαση αυτή, πολλοί αξιωματούχοι του Σοβιετικής Ένωσης και τώρα πολίτες της Ρωσικής ε, Ομοσπονδίας, ε, της Ουκρανίας και της Λιθουανίας καταδικάστηκαν ε, ως ένοχοι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου κατά της ε, Λιθουανικής Δημοκρατίας. Ε, Πριτάνευση δικαιοσύνη. Πέρυσι όμω η Εξεταστική Επιτροπή τη Ρωσική Ομοσπονδία εκείνησε ποινικέ διώξει κατά των ε, Λιθουανών εισαγγελέων που ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση και τον Απρίλιο ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του, των δικαστών που δίκασαν, εκδίκασαν αυτή την υπόθεση. Και μάλιστα με βάση τα άρθρα του ποινικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που ουσιαστικά έφεραν αθώους σε ποινική δίκη στα πλαίσια μιας άδικης δίκης. Κάτι που είναι πρωτοφανές και ανεφρεγουμένο και βάλει ανεπανόρθωτα κατά της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας Τη δικαστική εξουσία. Θεωρούμε τέτοιε δράσει της Ρωσικής Ομοσπονδία ως ε, ασύμβατες με το κράτος δικαίου και αξιοθρύνητε. Είναι απαράδεκτο να διώκονται δικαστές και εισαγγελεί μιας ανεξάρτητης χώρας μόνο και μόνο επειδή άσκησαν το συνταγματικό τους καθήκον και απένιμαν δικαιοσύνη τέτοιες δράσεις ε, στρέφονται κατά της ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και πλήττουν ε, τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Δικαστές μιας χώρας μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εισαγγελεί Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θύματα αυτής τη κατάστασης και δεν παραβιάζεται έτσι το κράτος δικαίου μόνο της Λιθουανίας αλλά του συνόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζεται και απειλείται άμεσα από τις δράσεις μιας τρίτης χώρας αυτή ήταν ε, μια επίθεση όχι κατά μόνο των λιθώνων δικαστών και εισαγγελέων, αλλά επίθεση κατά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, προβληματιζόμαστε ιδιαίτερως ε, με τη συνέπειε τη δράση τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θεωρούμε ότι είναι κατάχρηση των διμερών και πολυμερών συμφωνιών και κατάχρηση των διατάξεων για την έτσι έκδοση δικαστών και εισαγγελέων μετά από δίκη που είχε πολιτικά κίνητρα. Πιστεύουμε ότι η ελευθερία τους μπορεί να δεθεί σε κίνδυνο. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 19 Σεπτεμβρίου του 2019 με θέμα τη σημασία της ιστορική ε, μνήμη ιστορικής ε, για το μέλλον τη Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατράνωσε την θέση του σε ό,τι αφορά τις απόπειρες του Ρώσου ηγέτη να ε, διαστρεβλώσει τα ιστορικά γεγονότα για τα εγκλήματα ε, της Σοβιετικής Ένωσης και επίσης ε, έχουν ολόκληρη εκστρατεία παραπληροφόρηση κατά της δημοκρατικής Ευρώπης με απόπειρα να τη διαιρέσουν, να τη διχάσουν. Επίσης θα πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτές τις επικίνδυνες δράσεις κατά του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε αυτή την κατάσταση. Αν μια τρίτη χώρα αναλαμβάνει τέτοιε δράσεις κατά λιθωνών δικαστών και εισαγγελέων, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο, καμία εγγύηση ότι μία άλλη μέρα παρόμοιες δράσεις θα ασκηθούν κατά δικαστού εισαγγελέα άλλης χώρας μέλους. Σήμερα οι Λιθουανοί δικαστές και εισαγγελείς έχουν γίνει στόχος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αύριο όμως θα μπορεί να είναι οι Ολλανδοί που διερευνούν το ατύχημα του Μαλαισιανού αεροσκάφους. Ε, μπορούν να είναι οι Πολωνοί που προσπαθούν να, να διαλευκάνουν το αεροπορικό δυστύχισμα του Σμόλενσκ το 2010. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πρόσφατο ψήφισμά του δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως μοντέλο ειρήνης και επανασυφιλίωσης ήταν μια ελεύθερη επιλογή των λόγων της Ευρώπης που δεσμεύθηκαν σε ένα κοινό μέλλον και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη ευθύνη να προωθήσει και να διαφυλάξει τη δημοκρατία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει τις εξουσίες του και θα διαμαρτυρηθεί και θα στυλιτεύσει, θα καταδικάσει τις δράσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά Λιθουανών δικαστών και εισαγγελέων. Και επίσης θα ζητήσουμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία ε, να καταπολεμήσει την ατιμορρησία και να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και όχι να απειλεί ε, Ευρωπαίους δικαστές και να επιτίθεται στο κράτος δικαίου. Ελπίζουμε να είναι ξεκάθαρη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υιοθετήσετε και ένα νέο ψήφισμα ε, για την σημερινή κατάσταση. Είναι γεγονό ότι σήμερα μια τρίτη χώρα ήδη προσπάθησε να επηρεάσει τι εκλογικέ διαδικασίε σε κάποια κράτη-μέλη. Και μάλιστα η σημερινή απόφαση θα. Η σημερινή απόφασή σα θα κρίνει αν θα επιτρέψουμε σε μια τρίτη χώρα να, να παρέμβει στο, δικαστικό, στο δικαστικό μα σύστημα και να το επηρεάσει. Σίγουρα πιστεύουμε ότι θα πρέ... ο κόσμο θα πρέπει να είναι πιο ειρηνικό αύριο, αλλά σήμερα θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση. Μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Ελπίζω ότι τα μέλη τη Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών θα προσπίσουν το κράτο δικαίου και δεν θα, ε, δεν θα επιτρέψουν σε καμία χώρα να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Δικαστική Τάξη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που μα επισημάνετε το θέμα αυτό και που μα παρουσιάσατε την υπόθεση αυτή με τις συνέπειες ε, που θα μπορούσε να έχει για το κράτος δικαίου και την προάσπιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα και κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και του κράτους δικαίου. Να συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό, αλλά καταρχάς Ο κύριος Ευάλωτο Βασίλη ε, έχει το λόγο, ο Γενικό Εισαγγελέα ε, της ε, Λιθουανική Δημοκρατίας και μετά ο κύριο Μέλιος Νέργκιου, που είναι ο επικεφαλής του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Λιθουανία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Χαίρομαι που έχω το λόγο και είναι τιμή μου που μπορώ να σας μιλήσω. Ε, τα περιστατικά της του 1991 αφορούν τον α, ε, Υπουργό δικαιοσύνης, τον Υπουργό Ιστορικών και των ε, παραστατικών ομάδων. Τα εγκλήματα που διαπράχθησαν ε, περιλάμβαναν εκρηκτικούς μηχανισμούς, όπλα που οδήγησαν στην τη ζωή 14 ε, ατόμων αμάχων και στον τραυματισμό 800 ατόμων. Εμείς οι εισαγγελείς ε, εξετάσαμε και διαβάσαμε πάνω από χίλιες σελίδες σημαντικών τέτοιων ε, γράφων. Είδαμε χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες. Ανακρίναμε πάνω από 5.000 άτομα και λάβαμε και αποστήλαμε μάλλον 300 αιτήματα νομικής αρρωγής σε, σε άλλες χώρες και παρά το γεγονός ότι οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας αρνήθηκαν να συνεργαστούν στην προκειμένη περίπτωση, οι αρχές της Λιθουανίας α, ε, κυνήγησαν την υπόθεση αυτή και συνέλεξαν στοιχεία κατά 64 ατόμων Και αυτά ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 2019. Οι αρχές της Ρωσικής ε, Ομοσπονδίας έλαβαν συγκεκριμένα μέτρα για να φοβήσουν, εκφοβήσουν ε, ε, πολλούς στη Λιθουανία, τους δικαστές, τους εισαγγελείς. Επίσης, η παράνομα αυτή δίωξη επιβεβαιώθηκε σε σχέση με διάφορε ε, αιτήματα που έλαβαν ε, οι αρχέ της Λιθουανίας ε, το 2019. Η έρευνα γίνεται μαζί με μια επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την παράνομη αυτή δίωξη των πολιτών όπως προβλέπεται στο άρθρο 299 του ποινικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρόκειται για μέλη της Αγγελίας, της Λιθουανίας και δικαστές του Περιφερειακού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου του Μπελνίου το 2016 έγινε ποινική δίωξη των αξιωματούχων αυτών και διάφορα άτομα καταδικάστηκαν και τα οποία είχαν αναγνωριστεί από τις ρωσικές αρχές ως θύματα. Το άρθρο λοιπόν αυτό το 299 του ποινικού κώδικα προβλέπει στις φυλάκισης 5-10 ετών σε ό,τι αφορά τις ε, καταστάσεις που αποκαλύφθηκαν για τη Λιθουανία. Οι ποινικέ διώξεις που σχετίζονται με τις δράσεις των μυστικών υπηρεσιών στη Λιθουανία και σύμφωνα με τα στοιχεία που λάβαμε, τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν με την έρευνα κατά των Λιθουανών εισαγγελέων και δικαστών και αναφέρονται από τις αρχές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είναι βασικό να ληφθούν όλα τα μέτρα για να προστατευτούν οι δικαστέ και εισαγγελεί τη Λιθουανία. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι όταν η κατάσταση αξιολογηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βρεθεί μια σωστή λύση θα αποτελέσει μια βασική α, συμβολή για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματο στο ιστορικό και στο εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε και την κυρία Μελούτη, αλλά παρακαλώ. Έχετε τρία λεπτά κατά ανώτατο όριο για να υπάρχει και περιθώριο συζήτηση, ε, γιατί θέλουν να κάνουν οι βουλευτέ ερωτήσει προ τον ε, Υπουργό. Αξιότιμε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον της αξιότιμης επιτροπής σας. Συμφωνώ απόλυτα αυτά που είπε ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Δεν θα επαναλάβω όμω τα όσα είπε. Ωστόσο, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιε πτυχέ του θέματο, οι οποίε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικέ. Καταρχά, πιστεύω ακράδαντα. Πιστεύω ότι οι ρωσικές δηλώσεις για τις ε, έρευνες πρώτης ε, κατά των ε, Λιθουανών δικαστών και εισαγγελέων έχει πολιτικό υπόβαθρο και όχι τεχνικό νομικό υπόβαθρο. Θα σας πω ότι οι δικαστές οι οποίοι ήδη έχουν εκδώσει αποφάσεις και αυτοί που θα αποφανθούν για το θέμα αυτό σε επίπεδο εφετείου και ανώτατου δικαστηρίου. Οι δικαστές όμως δεν το έχουν κάνει αυτό, γιατί έχουν γίνει 15 αιτήματα, 15 εφέσεις. Άρα η ποινική διαδικασία είναι ακόμα ανοιχτή. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο για μα είναι τι θέλει να πετύχει η Ρωσία με τη δήλωση αυτή. Η Ρωσία έστειλε ένα πολύ απλό μήνυμα προ του δικαστέ. Να φοβούμαστε, να φοβούνται, γιατί θα του διώξουν. Αυτό προφανώ θα έχει αντίκτυπο στο δικαστικό σώμα. Είναι σαφέ προ όλου ότι οποιοδήποτε άτομο και οποιαδήποτε οργάνωση ή οποιοδήποτε κράτο έχει πλέον δικαίωμα να παρέμβει στο δικαστικό σώμα, στην ανεξαρτησία ενός άλλου κράτους. Επίσης, τέτοιες δηλώσεις σχετίζονται με την βασική και θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος δικαίου κατ' ουσίαν. Εμείς ως δικαστές λοιπόν έχουμε ακολουθήσει αυτή την βασική αξία και τα άλλα κρατημέλη επίσης υποστηρίζουν και προσπίσονται αυτή την βασική αξία τη θεμελιώδη αξία του κράτους δικαίου. Άρα ζητούμε όχι μόνο να ε, υπερασπιστούμε του ε, δικαστέ τη Λιθουανία, αλλά να επιβεβαιώσουμε ότι η Ευρώπη ακολουθεί την αρχή του κράτους δικαίου και να καταδικάσουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στην ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Το δεύτερο σημαντικό σημείο το οποίο θεωρώ ότι υπάρχει από πλευρά ε, του δικαστικού σώματος είναι ότι έχουμε λάβει δράση για να προστατεύσουμε τους δικαστές μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προτού λάβουμε και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Δικαστικό Συμβούλιο της Λιθουανίας ε, καταδίκασε δημόσια τέτοιες δράσεις της ε, Ρωσίας και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη. Και λάβαμε υποστήριξη λοιπόν από τι αρχέ μα. Ε, το Λουθενικό Συμβούλιο επίση ε, παρουσίασε την υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENCJ, το οποίο περιλαμβάνει και τα δικαστικά σώματα των ε, άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση. Συντήθηκε λοιπόν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ECJ το θέμα αυτό και επίσης μας υποστήριξε το δίκτυο αυτό επίσημα και δημόσια. Ωστόσο, Θεωρείτε ότι αυτό είχε οποιοδήποτε αντίκτυπο στη Ρωσία. Όχι, προφανώς αυτή είναι η απάντηση. Αυτό ε, επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία δεν ε, εισακούει οποιοδήποτε νομικό επιχείρημα, είτε από εθνικά, είτε από διεθνή σώματα και οργανώσεις. Και αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα εκ νέου ότι το θέμα αυτό είναι αμυγός πολιτικό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί πολιτικά με σαφήνεια σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή και να υπερασπιστεί τους δικαστές και προφανώς αυτό θα πρέπει να εκφραστεί και σε ένα ψήφισμα το οποίο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να υλοποιήσετε. Και τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε ό,τι αφορά την πράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Είναι η πρώτη τέτοια σοβαρή απόπειρα παρέμβαση σε ανεξάρτητα δικαστικά σώματα ένα κράτο μέλου. Αν δεν βάλουμε λοιπόν τώρα ένα τέρμα, αν δεν πούμε τώρα ω εδώ, δεν θα είναι η τελευταία απόπειρα αυτή. Αν ε, ανεχτούμε αυτή την απόπειρα παρέμβαση, τα αποτελέσματα θα είναι δραματικά. Αυτό θέλω λοιπόν να το λάβετε υπόψη του λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω την υπόθεση των Λιθουανών δικαστών ενώπιον τη Επιτροπή σα και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ήδη μια πρώτη μικρή νίκη για την προάσπιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος της Λιθουανίας. Αλλά παράλληλα ελπίζω να μην περιοριστεί η συζήτηση στην Επιτροπή σας, να το θέσετε το θέμα αυτό σε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο θα επιβεβαιώσει τη σημασία της αξίας του κράτους δικαίου, αλλά και θα προσπιστεί την εξαρτησία όλων των Ευρωπαίων δικαστών και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να μην με Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, να κάνουμε τη συζητήση και μετά θα σχολιάσει ο υπουργό τα όσα ακούσει. Βλέπω ότι έχετε σηκώσει τις κάρτες σας. Οι συντονιστές μπορούν να πάρουν πρώτο το λόγο, αν δεν το επιθυμούν, να δώσουν το λόγο κατευθείαν στην κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω και εσάς, Υπουργέ, για την πολύ σημαντική αυτή η παρέμβασή σα Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να πω ότι εξ ονόματο τη ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζουμε την Λιθουανία. Η σφαγή του 1991 είχε ε, μεγάλο αντίκτυπο που ξεπέρασαν τα σύνορα τη Λιθουανία. Αυτό το επεισόδιο το αντιλαμβάνεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι οι δικαστές της Λιθουανίας είναι Ευρωπαίοι δικαστές και θα ήθελα να τράξω την ευκαιρία για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στην προστασία των εισαγγελέων και των δικαστών της ε, Λιθουανίας που συμμετέχουν στις έρευνες για τα τραγικά γεγονότα της του 1991 στο Πελνίους. Είναι λοιπόν ανακριτέ και εισαγγελεί και δικαστέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να του προστατεύσουμε από παράνομε απόπειρε παρέμβαση από το εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Και θα να είστε βέβαιοι ότι η Λιθουανία θα δει ότι η ομάδα μας ε, και το κοινοβούλιο ολόκληρο θα τους υποστηρίξει. Είμαστε όλοι υπέρ λοιπόν του ανεξάρτητου δικαστικού σώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα έχει την, το δικαίωμα άσκηση των κατα τα τους εμ, χωρίς εξωτερικές επιρροές. Αυτό λοιπόν θα συζητηθεί σε όλες τις πολιτικές ομάδες, σε όλα τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι και του άνατο το επίπεδο να χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σίπελ, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτήν την παρουσίαση σήμερα και νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε την κατάσταση γιατί εδώ πέρα γύρονται δικαστικά ερωτήματα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αλλά βεβαίως σχετίζεται και με τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες και με την ε, λεπτή κατάσταση που υπάρχει ακόμα στην χώρα σας και τις ε, άλλες χώρες που συνορεύουν με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί να δούμε την κατάσταση, αλλά σαφώς πρέπει να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνη και των δικαστών όταν κάνουν την δουλειά τους σύμφωνα με τον νόμο. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό έχοντας κατά νου ότι όλα αυτά έχουν και μία εξωτερική πτυχή και θα πρέπει να γίνει μία ευρύτερη συζήτηση για να παρακολουθήσουμε και τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Λοιπόν, σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αρχή για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να δούμε το τι θα γίνει από εδώ και μπρος και πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε το δικαστικό μας σύστημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ίνετφελ, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Υπουργό και τους άλλους ομιλητές και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την στήριξή μου γιατί όπως σωστά είπατε οι Λιθουανοί δικαστές ε, και εισαγγελείς είναι Ευρωπαίοι δικαστές και οι εισαγγελείς. Δεν είναι διμερές το ζήτημα λοιπόν. Είναι θέμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της Ρωσίας και πρέπει να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα του δικαστικού συστήματος. Έχω κάποιες ερωτήσεις, γιατί δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Αν κατάλαβα καλά, αναφέρατε ότι αυτό έχει συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλίων Δικαιοσύνης και έχει υπάρξει κάποια καταδίκη. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Μετά μια ερώτηση προς ε, την Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να δούμε το τι συνέπειες θα έχει μια τέτοια κίνηση για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία με την Ρωσία. Δίνουμε προσωπικά δεδομένα, αστυνομικά δεδομένα στην Ρωσία. Θα μπορούσαν αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν κατά όχι μόνο οποιονδήποτε Ευρωπαίων πολιτών, αλλά δικαστών και εισαγγελέων. Τι σημαίνει αυτό. τι θα γίνει αν ε, ε, δοθούν τα νόματα αυτά στην Interpol. Πρακτικά τι σημαίνει. Τι αυτά είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να τους εκφοβήσουν. Πρώτα απ' όλα τι σημαίνει αυτό Λοιπόν, όχι να το ξαναπώ. Είναι ανοιχτή αυτή η υπόθεση. Πέρα από τις πολιτικές δηλώσεις, ε, νομικά τι μπορεί να γίνει. Παραδείγματος χάρη. Υπάρχει το δικαστήριο του Στρασβούργου. Τι άλλα νομικά μέσα έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι ε, η νομική οδός είναι πολύ πιο δύσκολη από το να κάνουμε κάτι πολιτικά και να πούμε ότι δεχόμαστε εκφοβισμό από τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ κυρία Ινετφέλντ. Τώρα κύριος Μπράιερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίασή σας και σας διαβεβαιώ πως ε, και η δική μου ομάδα, η πράσινη, ε, είμαστε αλληλέγγυοι γιατί βεβαίως η αρχή της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα πέρα από αυτό το συγκεκριμένο το οποίο λέτε, ανησυχούμε κάπως γενικότερα για την πολιτική χρήση κάποιων μέσων. Αυτό ισχύει παραδείγματο χάρη για το μηχανισμό της Interpol που φαίνεται ότι ε, χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για πολιτικές διώξεις. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τα κράτη-μέλη που εκτελούν ε, εντάλματα σύλληψης ατόμων που εντάλματα που έχουν εκδοθεί για πολιτικούς λόγους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και στην δική σας περίπτωση. Και υπάρχει αυτό το οποίο είπε η κυρία Ινέτφελντ. Έχω μια ερώτηση λοιπόν. Έχετε ενδείξεις για το ότι δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούνται στην έρευνα αυτή στη Ρωσία γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε γενικότερα. Μην ε, βοηθάμε τέτοιες διαδικασίες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία είναι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε το θέμα. Θα μιλήσω την Λιθουανική και από κάποια γενικότερα πράγματα. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε την περίπτωση αυτή στο γενικότερο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου που διεξάγει το Κρεμλίνο. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι το διάδοχο κράτος της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά ένα στόχος του Κρεμλίνου είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει νομικό ηθικό αίρεσμα για τα σοβιετικά εγκλήματα, οπότε εδώ πέρα υπάρχει πλήρης άρνηση της κατοχής ε, της ε, Λιθουανίας. Υπάρχουν προσπάθειες για να μην φροντίσουμε τα νεκροταφεία των εκτοπισμένων. Αυτά τα κάνει η Ρωσία και κατά των ίδιων των πολιτών της, αλλά για πρώτη φορά ασκεί η πολιτική τρομοκρατία κατά δίκαστων και εισαγγελέων σε άλλη χώρα. Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο, όπως είπα, για να εκδικηθεί για τις καταδίκες αυτές και είναι μια προσπάθεια για να επηρεάσει και τις μελλοντικέ αποφάσεις. Αν η Ρωσία δεν λάβει μια σαφή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι τελείως απαράδεκτο αυτό, τότε και άλλοι δικαστές και εισαγγελείς που εργάζονται σε οποιαδήποτε υπόθεση θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο εάν το Κρεμλίνο αρνείται τις ε, ευθύνες του. Ας δούμε την πτήση MH70, την κατάρριψή της. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε μία ακρόαση όπου θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα από τέτοιες παρεμβάσεις και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό να απαντήσει γιατί θα είναι σημαντικό ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. The Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ήμουν από τους μάρτυρες των γεγονότων της 13ης ε, Ιανουαρίου του 1991. Ήμουν τότε υπουργό Υγεία και είδα τους τραυματισμένους και δολοφονηθέντες συμπολίτε μου. Ήταν τραγική αυτή η περίπτωση, αλλά σήμερα δεν συζητούμε τα τραγικά γεγονότα του Ιανουαρίου του 1991, αλλά το κράτος δικαίου και την κατάσταση Ευρωπαίων δικαστών και Εισαγγελίων που έκαναν το καθήκον τους έλαβαν μία απόφαση και εξέδωσαν μία απόφαση ε, κατά, μίας, ε, κατά πολιτών τρίτης χώρας και αυτή η τρίτη χώρα άσκησε ποινικέ διώξεις κατά Ευρωπαίων δικαστών και εισαγγελίων. Γι' αυτό ε, φέρνουμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τον Υπουργό, τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου του Κάουνας που μας παρουσίασαν την περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την υπόθεση για να μην δημιουργηθεί προηγούμενο παρέμβαση μιας τρίτης χώρας στην, στο κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συντάξουμε ψήφισμα στυλιτεύοντας αυτή την παρέμβαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι και η πρώτη, είχαμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ συμφωνώ με τον Υπουργό και πιστεύω ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συντάξει σχετικό ψήφισμα με τη θέση του. Αυτό θα το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θα εκπονήσει ένα τέτοιο ψήφισμα, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα και πολύ φόρτο εργασίας Πάντως αν υπάρχει βούληση και αν το συμφωνήσουν οι συντονιστές, θα ακολουθήσουμε τις, κανονικ... τις ε, συνήθες διάβλους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρίνει ένα σκόπιμο να σε ένα τέτοιο ψήφισμα. Πάντως νομίζω ότι δώσαμε την προσοχή της άξης στην υπόθεση αυτή, γιατί πραγματικά επηρεάζει τη... την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που είναι από τις ιδρυτικές αρχές και αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θεμελιώδη ζήτημα κράτους δικαίου, η προστασία της ανεξαρτησίας των δικαστών και εισαγγελέων, ε, ιδιαίτερα όταν ε, εκδικάζουν ποινικέ υποθέσεις και όταν ε, ε, ερευνούν ή απαγγέλουν κατηγορίες ε, κατά δραστών εγκλημάτων που θίγουν τα θεμέλια και τις ε, θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα ξαναδώσω το λόγο στον Υπουργό για να ολοκληρώσουμε. Θα μιλήσω λιθουανικά τώρα. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ευχαριστώ κυρία Μέτσολα, κυρία Τσίβελ, κυρία Χίντβελ, κύριε Μπράιερ για την υποστήριξή σας. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ενότητα και Αλληλεγγύη και μας ενδιαφέρει και η προβολή αυτού του θέματος και χαίρομαι που όλοι αντιληφθήκατε ότι οι Λιθουανοί δικαστές και εισαγγελείς είναι Ευρωπαίοι δικαστές και εισαγγελείς που χρήζουν και αξίζουν προστασίας. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Ιντβελτ ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ο δικαστικό Συμβουλίων ε, εξέτασε το θέμα και θα πρέσει την υποστήριξή του προς τους λιθόνους δικαστές και μάλιστα υπέβαλε και σημείωμα προς την Επιτροπή σας. Τι θα γίνει στη χειρότερη περίπτωση για αυτούς τους λιθόνους ε, δικαστές και εισαγγελείς που διώκονται. Φανταστείτε ένα σενάριο που δικαστές και εισαγγελείς ε, μπορεί να ταξιδέψουν σε τρίτες χώρες, μπορεί και να συλληφθούν και άρα να παραβιαστεί η ελευθερία τους. Έχουμε και το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Δεν θα επεκταθώ στο θέμα αυτό. Πάντως μια σύντομη απάντηση θα ήταν ότι ναι, χρησιμοποιούνται δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση αυτή. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευκαιρία που μου δώσετε να σας παρουσιάσω την κατάσταση και ελπίζω ότι η Επιτροπή σας θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την εκπόνηση σχετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και τους Λιθουανούς Ευρωβουλευτές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κύριε Μπράουρ, έχετε κάποια συμπληρωματική παρατήρηση. Άλλωστε πρέπει να ξαναδώσω και πάλι το λόγο στον Υπουργό. Ναι, θα συνεχίσω αυτά που είπατε. Είπατε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά δεδομένα κατά την άσκηση αυτών των διώξεων κατά των Λιθουανών δικαστών. Σας κατάλαβα καλά. Ε, τη χρήση τέτοιων δεδομένων από πλευράς Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν είμαστε βέβαιοι. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για μια πολιτική αξιολόγηση της υπόθεσης. Για την έκφραση μιας πολιτικής κρίσης δηλαδή της Επιτροπής μας. Ε, Υπάρχουν όλα τα στοιχεία για ανάληψη πολιτικής δράσης και από πλευράς Επιτροπής και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως χαίρομαι που ακούσαμε την παρουσίαση της υπόθεσης αυτής από ένα κράτος μέλος που τάσεται υπέρ της προστασίας της δικαστικής εξουσίας ενός κράτους μέλους και ευχαριστούμε τον Λιθουανό Υπουργό δικαιοσύνης για την παρουσίαση που μας έκανε της υπόθεσης αυτής. Έχω όμως και ένα άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το τελευταίο, που αφορά το ενημερωτικό έγγραφο του ελεκτικού συνεδρίου. Ευχαριστούμε ε, τον Λιθουανό Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Λιθουανό Γενικό Εισαγγελέα και τον εκπρόσωπο του Περιφερειακού Δικαστικού Συμβουλίου που ήρθαν εδώ και μας παρουσίασαν την υπόθεση αυτή. Λοιπόν, συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που έμειναν και κάποιοι στην αίθουσα. Οπότε έχουμε τα δύο τελευταία σημεία της ημερησίας διάταξης, στα οποία θα προεδρεύσω εγώ. Γιατί ο Χουάν Φερνάντο είχε άλλες υποχρεώσεις. Το επόμενο σημείο λοιπόν αφορά την ενημέρωση από το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο λέγεται «Προκλήσεις αποτελεσματικής πολιτικής κυβερνοασφάλειας». Και παρακολουθούμε το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής των υπηρεσιών των αρμοδίων και της ε, Κομισιόν. Και αυτό το οποίο ενδιαφέρει την Επιτροπή μας, πέρα από την ε, νομιμότητα το και την κανονικότητα των δαπανών είναι και οι ενημερώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που εξετάζει την απόδοση των πολιτικών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον κύριο Τομέ ο οποίος ε, θα μας ε, παρουσιάσει το έγγραφο αυτό και μετά θα δώσω τον λόγο στους βουλευτές. Κύριε Τωμά, έχετε τον λόγο. Thank you, Madam Chair. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που μου δίνετε ευκαιρία να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας το ενημερωτικό έγγραφο που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο τον περασμένο Μάρτιο στο οποίο παρέχουμε μια ευρή επισκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιτύχει μια αποτελεσματική πολιτική για την κυβερνοασφάλεια. Το ελεκτικό συνέδριο επεκτείνεται σε νέους τομείς ε, και νέες αρμοδιότητες, ακολουθώντας τις δραστηριότητες και προτεραιότητες της Ένωσης. Πρόσφατα ε, χρειάστηκε να συστήσουμε μια ειδικευμένη ομάδα ελεγκτών προκειμένου να ελέγξουμε θέματα συναφή με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και την νέα οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα τομέα καινούριο για μα, πρωτόγνωρο και χρειάστηκε να επεκταθούμε και σε αυτόν. Σήμερα ξεκινάμε την ενασχόληση με θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα τομείς που είναι πολύ σημαντικοί και έχουν προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ε, και το Ελεκτικό Συνέδριο και τα άλλα θεσμικά όργανα χρειάστηκε να επεκταθούν και σε αυτούς τους τομείς, αναλαμβάνοντας νέες προκλήσεις. Στα πλαίσια του ενημερωτικού αυτού εγγράφου θα ήθελα να σας κάνω μια παρουσίαση και να σας παραπέμψω επίσης στην ανάλυση απαριθμών 9 του 2019 με θέμα την Ευρωπαϊκή Άμυνα. ή πρόσφατες ε, εκθέσεις που έχουμε δημοσιεύσει με θέμα τον έλεγχο των συνόρων ή τα συστήματα πληροφορικής για θέματα ελευθεριών και ελέγχου των συνόρων. Το ενημερωτικό έγγραφο που θα σας παρουσιάσω σήμερα δεν είναι ένα άμυγες έγγραφο ελέγχου. Ουσιαστικά κάνει μια επισκόπηση των θεμάτων ε, και των εκθέσεων που έχουμε συγκεντρώσει προκειμένου να ετοιμάσουμε τις μελλοντικές μας εκθέσεις ε, με περιεχόμενο ελεκτικό και που αναμένονται με ενδιαφέρον από τους ε, εμπλεκόμενους φορείς. Για να υλοποιήσουμε αυτό το έγγραφο έχουμε χρησιμοποιήσει δημόσια έγγραφα, συνεντεύξεις, εκθέσεις και αναλύσεις από διάφορες πηγές. Ε, επίσης χρησιμοποίησαμε και μία έρευνα, μία, ένα ερωτηματολόγιο μάλλον, που στείλαμε στους ανώτατους ελεκτικούς φορείς των κρατών μελών για να απαντήσουν. Όπως ξέρετε, η κυβερνοασφάλιση είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στους σημερινούς καιρούς καθημερινά χρησιμοποιούμε περισσότερη τεχνολογία και είμαστε όλο και πιο ευάλωτοι απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις. Ως εκ τούτου η κυβερνοασφάλεια είναι κάτι που ενδιαφέρει πια άμεσα και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Με το ενημερωτικό αυτό έγγραφο εξετάσαμε το πολυσύνθετο τομέα της κυβερνοασφάλειας και εντοπίσαμε 10 σημαντικές προκλήσεις που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε τέσσερις κατηγορίε. Καταρχήν, το πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο, δεύτερον, δημόσιες δαπάνες και χρηματοδότησή τους, τρίτον, ενίσχυση της κυβερνοαθεκτικότητας και τέταρτος, τέταρτη κατηγορία, αποτελεσματική αντιμετώπιση των κυβερνοπεριστατικών, των περιστατικών της κυβερνοασφάλειας. Στα πλαίσια του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το περίπλοκο οικοσύστημα του κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αλληλεπίδραση πολλαπλών φορέων και παραγόντων. Και γι' αυτό ακόμη και η διαμόρφωση μιας γενικής θεώρησης όλων αυτών των οργανισμών, των θεσμών, των φορέων, των επιτροπών στα κράτη-μέλη και μόνο μια τέτοια γενική θεώρηση είναι ήδη μεγάλη πρόκληση λόγω του πολύ σύνθετου τοπίου. Νομίζω όμως ότι κάναμε μια επισκόπηση που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στους ενδιαφερόμενους. Στο πρώτο παράρτημα μάλιστα της έκθεσής μας, του ενημερωτικού εγγράφου μας, βλέπετε πόσο περίπλοκο είναι το πανόραμα που αναλύσαμε, το τοπίο που αναλύσαμε. Άλλο, άλλη σημαντική πρόκληση ε, είναι η αξιολόγηση και η ποσοτικοποίηση, η αποτελεσματική ποσοτικοποίηση των συνοποιών των δράσεων που έχουν αναλυθεί, προκειμένου να, ε, να εγγυηθούμε μία άρτια λογοδοσία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ποσοτικοποιημένους στόχους και έγκυρα στοιχεία. Επίσης, ε, ε, το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι ατελές και κατακαιρματισμένο και δεν έχουμε απόλυτη συνοχή στη μεταφορά των νομοθετικών ε, διατάξεων στα κράτη-μέλη, όλα αυτά εμποδίζουν την αξιοποίηση στο έπακρο του νομοθετικού πλαισίου. Επίσης, ε, θα πρέπει οι νομοθέτες ε, να προλαμβάνουν τις μελλοντικές εξελίξεις, ώστε στο μέτρο που εξελίσσεται ραγδαία η τεχνολογία και οι κυβερνοαπειλές, να μπορούμε και εμείς να δώσουμε μια αποτελεσματική απάντηση σε όλα αυτά και να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υλοποιήσει το στόχο να γίνει ο πιο ασφαλής ψηφιακός χώρος του κόσμου, θα πρέπει να αντιμετωπίσει προκλήσεις και σε επίπεδο δαπανών και άρα να καταβάλει σημαντικές ε, δημοσιονομικές προσπάθειες. Θα πρέπει επίσης να προσαρμόσει τα επίπεδα επενδύσεων στους στόχους που θέλει να υλοποιήσει. Κάτι που προϋποθέτει αύξηση όχι μόνο των ε, συνολικών επενδύσεων στην κυβερνοασφάλεια που μέχρι στιγμή ήταν περιορισμένες και κατακαιρματισμένες και αποσπασματικές. Θα πρέπει ταυτόχρονα να βελτιώσουμε τις ε, επιπτώσεις αυτών των επενδύσεων αξιοποιώντας καλύτερα τα αποτελέσματα των δαπανών στην έρευνα, εξασφαλίζοντας καλύτερη επιλογή και χρηματοδότηση των ε, σχεδίων και προγραμμάτων των αναφιωμένων επιχειρήσεων των αναδιαμένων επιχειρήσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε μια ξεκάθαρη γενική θεώρηση των δαπανών της Ένωσης και των κρατών μελών για να ε, γεφυρώσουμε πιθανές αδυναμίες. Το γεγονός ότι ε, έχουμε ένα ειδικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια ε, το, το γεγονό μάλλον ότι δεν έχουμε τέτοιο ξεκάθαρο προπολογισμό, ειδικό προπολογισμό τη Ένωση, δεν μα επιτρέπει να έχουμε σαφή άποψη για το, το επίπεδο και τον τρόπο των επενδύσεων και των δαπανών. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα τη κυβερνοασφάλεια να το δούμε οριζόντια. Επίση, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στην ανάγκη ε, εξασφάλιση απαραίτητων πόρων για του Ευρωπαϊκού Οργανισμού που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια, τον ΕΝΙΣΑ, την Europol, το CERT, EU. Αυτός, αυτή είναι μια πολύ περίπλοκη πρόκληση και ακριβώς η προσέλκυση ταλέντων και το, το να κρατήσουμε τα ταλέντα αυτά και το ανθρώπινο δυναμικό στους οργανισμούς είναι πολύ σημαντικό. Για να υλοποιήσουμε λοιπόν το στόχο της κυβερνοαθεκτικής κοινωνίας, θα πρέπει να διορθώσουμε τα κενά στη διακυβέρνηση της κυβερνοασφάλεια που εντοπίζονται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό κλάδο. Η διακυβέρνηση της κυβερνοασφάλεια συνίσταται στη διαχείριση των απειλών και των κινδύνων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων, σε μια σωστή ευαισθητοποίηση, καθώς και έναν σωστό συντονισμό και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ένα άρτιο μοντέλο διακυβέρνησης επηρεάζει σίγουρα την ικανότητα αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων και της του περιορισμού των κυβερνοεπιθέσεων. Γι' αυτό έχει κύρια σημασία να βελτιώσουμε τις ικανότητες και την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών μας. Η παιδεία, η εκπαίδευση λοιπόν και η κατάρτιση θα είναι σημαντικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας. Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αμοιβές εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων φορέων που ενεργοποιούνται στον τομέα της παγκόσμιας κυβερνοασφάλειας που είναι πολύ και διάφοροι και εμφανίζονται σε διάφορα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο γενικό συντονισμό είναι ανεπαρκής. Οπότε θα πρέπει να βελτιωθεί και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Κάποιες επιχειρήσει ήταν ιδιαίτερα πρόθυμε στο να μοιραστούν πληροφορίε για κυβερνοεπιθέσει ή κενά στην ασφάλειά του για να μην επηρεαστεί το κύρος του. Κάτι που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Γι' αυτό η βελτίωση τη ανταλλαγή πληροφοριών και η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα εξακολουθούν να συνιστούν σημαντική πρόκληση. Παρά τις ε, δράσεις που έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής, τα ψηφιακά συστήματα είναι τόσο περίπλοκα, ώστε η πρόληψη όλων των ε, επιθέσεων είναι ανέφικτη. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, αποτελεσματικά τα διάφορα περιστατικά και γι' αυτό Απαιτείται έγκαιρη, έγκαιρος, εντοπισμός και άμεση αντίδραση. Κάτι που προποθέτει καλό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των κοινωτικών θεσμικών οργάνων, καθώς και μια συντονισμένη διαχείριση των κρίσεων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προστατεύσουμε κατάλληλα τις κρίσιμες υποδομές και τις βασικές κοινωνικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, είχαμε τις πιθανές παρεμβάσεις, εκλογικές διαδικασίες ή τις εκστρατείες παραπληροφόρησης. Στο συγκεκριμένο ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου θα βρείτε πολύ πιο σχολαστική και διεξοδική ανάλυση που πραγματοποίησε το Ελεκτικό Συνέδριο σε όλους αυτούς τους τομείς και τις προτεραιότητες που σας παρουσίασα. Θα ήθελα εν κατακλείδη να επισημάνω ότι παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έκαναν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των κυβερνοαπειλών, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή ε, και απαραίτητη για να ενισχύσουμε την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή μας αυτονομία, χωρίς μάλιστα να διακυβεύσουμε τις θεμελιώδεις μας αξίες, που είναι η έμπνευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ενίσχυση της κυβερνοασφάλεια ε, θα απαιτήσει ε, προσοχή και αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων που αναφέραμε και θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, αξιολόγηση γεφυρώνοντας τα νομικά κενά που ίσως υπάρχουν. Θα πρέπει στη συνέχεια να αυξήσουμε τις επενδύσεις και να βελτιώσουμε τις συνέπειες και την αποτελεσματικότητά τους, να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση, τις ικανότητες και τις γνώσεις μας και να ενισχύσουμε ταυτόχρονα το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και επίσης να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική προστασία των κρίσιμων υποδομών και των βασικών ε, κοινωνικών λειτουργιών. Θα ήθελα εν τέλει να ευχαριστήσω την, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο, τους οργανισμούς ΕΝΙΣΑ και Ευρωπόλ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας και τους ανώτατους φορείς, ελεκτικούς φορείς των κρατών μελών για την, ε, για την ενθουσιώδη και επικοδομητική του συνεργασία και επίσης να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για το ενδιαφέρον που έδειξε ε, και ελπίζω το συγκεκριμένο ενημερωτικό έγγραφο και οι εκθέσεις μας ε, να είναι πηγή έμπνευσης ε, και να φανούν χρήσιμες στο έργο σας. Όπως είπα, χρησιμοποίησα, χρησιμοποίησαμε για τη σύνταξη του εγγράφου μας πολλοί άριθμες πηγές, φαίνονται και στη βιβλιογραφία, θα δείτε πάνω από 20 αναφορές εκθέσεων που να επαναλαμβάνω, τις ε, πηγές μας για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου. Είμαι στη διάθεσή σας και θα μπορούσα να απαντήσω στις απορίες σας ή να σχολιάσουμε ό,τι σας ενδιαφέρει σε σχέση με το έγγραφό μας. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ακούσαμε ήδη στην παρουσίασή σας αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για την ε, κυβερνοασφάλεια όχι μόνο στις υπηρεσίες αλλά και ως πρόκληση για τα κρατημέλη και είμαι ιδιαίτερο χαρούμενη για το ότι μιλήσατε για επενδύσεις σε διαφορούς ε, τομείς, για εκπαίδευση και ενημέρωση στο εθνικό επίπεδο. Βεβαίω μιλήσατε και για τον προϋπολογισμό, καθώς δεν υπάρχει σαφής ε, γραμμή στον προϋπολογισμό για το θέμα αυτό και χρειαζόμαστε και περισσότερα λεφτά. Ας δούμε τι θα κάνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Υπάρχουν πολλοί τομεί στους οποίους χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά ε, και ταυτόχρονα δεν ξέρω από πού θα μπορούσαμε να πάρουμε, ε, να ξοδέψουμε κάπου λιγότερα. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι στην ε, έκθεση αυτή ακούσαμε τόσα πολλά σημαντικά πράγματα. Σημαντικά για όλους μας. Κοιτάω Εάν κάποιος συνάδελφος να έχει κάποια ερώτηση. Ο κύριος εδώ πέρα, Πράιερ, είναι ο πρώτος συνάδελφος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που θίξατε το σημαντικό αυτό θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας που όπως είπατε δεν είναι προφανές αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ θετικό το ότι το εξετάζεται. Μάλιστα, με το ίντερνετ των πραγμάτων που έχουμε σήμερα, οι υπολογιστές επηρεάζουν τον κόσμο μας με τρόπο άμεσο και φυσικό, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, τα νοσοκομεία, οι ανασφαλείς ε, ηλεκτρονικές συσκευές ε, σημαίνει ότι μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή μας και η περιουσία μας. Δεν μπορούμε πλέον να βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοιες καταστροφές ε, καθημερινά. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά συνεχώς ε, βλέπουμε και υπάρχει μια έλλειψη ασφαλείας αυτή τη στιγμή. Η έκθεση σας βλέπω επίσης ε, δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο, άρα δεν ε, περιέχει τις τελευταίες εξελίξεις. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν κάποιες πτυχές για τις συμβάσεις για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που υπάρχει μια υποχρέωση για την παροχή ενημερώσεων ασφαλείας στους καταναλωτές. Υπάρχει επίσης ένα εθελοντικό σχέδιο πιστοποίησης, υπάρχει χρηματοδότηση για καλύτερη κυβερνοασφάλεια, όμως συμφωνώ ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι να είναι πιο σαφές για τους καταναλωτές ποιες ιδιότητες ασφαλείας έχουν τα προϊόντα. Βλέπουμε ένα προϊόν στο ράφι με στιγμής από την Κίνα ή από κάπου αλλού και δεν έχουμε ιδέα για το αν υπάρχουν αναβαθμίσεις, αν τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα, οι καταναλωτές δεν μπορούν να ξέρουν κάτι τέτοιο και δεν ξέρουν επαρκή επιστοποίηση. Μπορούσαμε να έχουμε κάποια διαφάνεια, κάποιο σύστημα σήμανσης των προϊόντων επίσης. Η αξιοπιστία των κατασκευαστών που δεν αντιδρούν όταν τους αναφέρουν κάποιες αδυναμίες. Ε, θα ήταν ένα κίνητρο νομίζω το να θεωρούνται υπεύθυνοι ε, για ζημιές αν δεν ε, διορθώνουν τα προβλήματα του λογισμικού τους. Επίσης πολλές αρχές προτιμούν να εκμεταλλεύονται αυτές τις ε, αδυναμίες για μέτρα παρακολούθησης αντί να τις κλείσουν. Και βεβαίω αυτό σημαίνει ότι τις αδυναμίες αυτές μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και οι εγκληματίες. Οπότε μια πολιτική του να κλείνουμε τις αδυναμίες αντί να τις εκμεταλλευόμαστε, τα βοηθούσε. Φοβάμαι όμως ότι η Europol κάνει το αντίθετο και έχει στήσει ένα φόρουμ για το πώς θα εκμεταλλευτεί αυτές τις πίσω πόρτες ε, του λογισμικού. Επιπλέον, όταν μιλάμε για κυβερνοεπιθέσεις, ε, η ανθεκτικότητα είναι πολύ πιο σημαντική από το να προσπαθήσουμε μετά να κάνουμε κάτι. Δηλαδή ο σχεδιασμός ε, των προϊόντων ε, εξ αρχής ώστε να μην ε, δέχονται επίθεση είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Από το να προσπαθούμε να εντοπίσουμε επιθέσεις που συχνά είναι αδύνατον. Τέλος, η έκθεσή σας μιλάει για το ζήτημα της διακράτησης δεδομένων και θα ήθελα να τονίσω ότι το ΔΕΚ ε, είπε ότι η γενική διακράτηση δεδομένων είναι δυσανάλογη και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και δεν εμποδίζει την αποτελεσματική δίωξη και αντιθέτως ε, τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν υποχρεωτική ε, διακράτηση δεδομένων όπως η Γερμανία ερευνούν τέτοια περιστατικά με εξίσου μεγάλη αποτελεσματικότητα με άλλες χώρες. Και δεν είχαμε δει επίσης ε, με την αντίθετη πολιτική κάποια αύξηση στην εξυχνίαση εγκλημάτων. Οπότε θα πρέπει να απορριφθεί αυτό το σκεπτικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπράιερ. Ε, είχατε την ευκαιρία αυτή και κάνατε πολλές ερωτήσεις. Ευτυχώς, γιατί φοβήθηκα ότι θα τελειώναμε. Δεν ε, ηρωνεύομαι. Λοιπόν, έχω κι άλλον ένα συνάδελφο. Ο κύριος Ασάλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την παρουσίαση. Είναι πολύ θετικό που το Ελεκτικό Συνέδριο ασχολείται και με το τόσο σημαντικό αυτό θέμα και μάλιστα υπό το πρίσμα του Ελεκτικού Συνεδρίου και από τη θέση που έχει το Ελεκτικό Συνέδριο στο όλο θεσμικό πλέσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ε, μας είπε ο κύριος Τομέ, το έγγραφο αυτό είναι ενημερωτικό και προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικούς ελέγχους. Δεν είναι καθ' αυτό έγγραφο ελέγχου. Ρωτώ λοιπόν, έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας με προτεραιότητες, με συγκεκριμένους τομείς ε, στους οποίους θα εγγύψει ελεκτικά πια το ελεκτικό συνέδριο. Και έρχομαι εδώ σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είστε υπέρα ενός ειδικού προϋπολογισμού ε, που θα αποτυπώνει την δημοσιονομική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια δεδομένης της οριζόντιας διάστασης που έχει αυτή η προσπάθεια. Κατάλαβα ότι μάλλον προτιμάτε ένα τέτοιο ειδικό προϋπολογισμό. Επίσης είπατε θα πρέπει να προκοδοτήσουμε επαρκώς τους διάφορους οργανισμούς της Ένωσης ε, που ασχολούνται με θέματα κυβερνοασφάλειας. Μιλούμε όμως για τι είδου ε, ε, εφόδια, οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό ή νομικούς μηχανισμούς και εργαλεία για την δράση τέτοιων οργανισμών. Σας ευχαριστώ. Να σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε σε όλα αυτά τα σχόλια και σε ερωτήσει. ερωτήσεις. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και το Καινούργιο Κοινοβούλιο αποδεικνύει με τη σχολιά της ότι η νέα μας αυτή η πρόταση έκθεση είναι ενδιαφέρουσα. Περιγράφονται λοιπόν πολλές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, του Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις γενικές διευθύνσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Και είναι σαφές ότι υπάρχουν, υπάρχει κίνηση και προφανώς υπάρχει και ευαισθητοποίηση και είναι πολλές οι που λαμβάνονται. Να αναφερθώ σε κάποιες από τις πτυχές τις οποίες επισημάνατε για την έκθεσή μας, για την ενημέρωσή μας. πιστοποίηση καταρχάς, μία από τις τελευταίες εξελίξεις που προέκυψαν από τον κανονισμό. εθελούσια συστήματα πιστοποίησης. Κόβεται δυστυχώς το μικρόφωνο του μιλτή. Σε ό,τι αφορά την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Αλλά σίγουρα η πιστοποίηση θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για τους μεγάλους παράγοντας ε, για μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, ε, συσκευές καταναλωτών, υπηρεσίες προς τον καταναλωτή. Φαντάζομαι ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι λειτουργεί η πιστοποίηση. Επίσης, Μιλήσατε για το διαδίκτυο των πραγμάτων και πώς εξελίσσεται. Νέες τεχνολογίες ανακύπτουν. Τα δίκτυα 5G. Θα μας επιτρέψουν να κάνουμε πιο εντατική χρήση των συσκευών IT. Θα προκύψουν και προκλήσεις προφανώς. θα έχουμε αποκεντρωμένα δίκτυα με μικρότερο έλεγχο. από τους ε, παραδοσιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιών. Προφανώς όσο επεκτείνεται το πεδίο μας τόσο πιο πολύ είναι κίνδυνοι. και παρακολουθούμε ενδεχόμενους κινδύνους που θα ανακύψουν. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εισαγωγέας τεχνολογίας, καθαρός στον τομέα αυτό. Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου μιλητής. You have referred... Um, ε, okay. You can... you have refer... Επίσης, αναφερθήκατε στο νομικό πλαίσιο για την ε, τήρηση δεδομένων. Δεν τοποθετούμαστε από αυτού. Εμείς Έχουμε συγκεράσει διάφορες πηγές πληροφοριών και έχουμε χαρτογραφήσει την κατάσταση όσο έχει. Αλλά, όντω, για την ε, καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος χρειάζεται ένας κάποιος συντονισμό. Και σε κάποιες περιπτώσεις, λοιπόν, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι εγκληματίες και πού και πώς βρουν. Υπάρχουν και αυτές οι υβριδικές απειλές. Ως τώρα δεν υπάρχει κάποιος συντονισμένος τρόπος ε, αντιμετώπισης των κινδύνων της κυβερνοασφάλειας. Χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω ανάλυση. Αυτό είναι σαφές από την έκθεσή μας για το πώς μπορούμε να καλύτερα την καταπολέμηση του κυβερνού Αν Αναφερθήκατε σε θέματα ανθεκτικότητας ευαισθητοποίησης και ένα από τα θέματα που αναφέραμε είναι και η εκπαίδευση, η κατάρτιση του κόσμου. Γιατί η αντίδραση είναι σημαντικός παράγοντας. Όλοι και οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και η αναφορά των κινδύνων και των απειλών είναι σημαντικό στοιχείο. Οι εταιρείε, ε, οι πάροχοι, οι εταιρείε ε, τηλεπικοινωνιών, οι αεροπορικές εταιρείε, οι σιδηροδρομικές εταιρείε, ε, μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις και μη που πρέπει να υποβάλουν αφορά για το τι συμβαίνει, αλλά για να προστατευτούν και οι ίδιες. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Δεν ξέρουμε πόσο επενδύονται στην κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προπολογισμό δεν είναι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και σε εθνικό επίπεδο. Και σε κάποιε περιπτώσει ο προπολογισμό αυτό δεν είναι αμυγό για την κυβερνοασφάλεια. Εξυπηρετεί και άλλου σκοπού. Έχουμε βρει κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τι ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι στι ΗΠΑ. δαπανάτε 0,3 του ΕΕΠ στην κυβερνή ασφάλεια. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Απέχουμε παρασάγκα από αυτά. I have together with me, ε, Έχω μαζί μου τον κύριο Μίχελ Σφέρτσα, ο οποίος είναι ο βασικός αρμόδιο από το ελληνικό συνέδριο για τέτοια θέματα και μπορεί να πάρει το λόγο, αν επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε. Ναι, έχουμε άλλα τρία λεπτά. Μήπω θέλετε να ολοκληρώσετε τη δική σα ομιλία. Και κύριο Αρθαλέχο. Ο κύριος Αρθαλέχος με ρώτησε για το πρόγραμμα εργασιών που έχει το ελεκτικό συνέδριο. Μετά την ανάλυση του θέματος βάζουμε στο πρόγραμμα και κάποιους ελέγχους που θα πραγματοποιήσουμε κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης που έχουν μεγάλη εμβέλεια. Επίσης, δράσεις των θεσμικών οργάνων, οργάνων για προστασία από διάφορες απειλές. Πάντως είναι ευρύτατο το πεδίο. Κάθε κεφάλαιο της έκθεσής μας καταλήγει σε ανοιχτές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να είναι πολύ ενδιαφέρουσες και στο επόμενο στάδιο το ελεγκτικό και θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τους ηθήνοντες πολιτικής και να τους βοηθήσουν στη χάραξη πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το κατά πόσο χρειαζόμαστε ειδικό προπολογισμό της Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια, εμάς μας ενδιαφέρει η ποσοτικοποίηση των δαπανών. Δεν έχει ίσως νόημα να έχουμε έναν ειδικό προϋπολογισμό για την κυβερνοασφάλεια. Γιατί η κυβερνοασφάλεια είναι οριζόντιο θέμα. Καλύπτει και τις ε, εξωτερικές δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπίπτει δηλαδή σε αυτή την παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά περιλαμβάνεται και στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Αγοράς για τα ψηφιακά θέματα. Οπότε θα υπάρχουν σχετικές δημοσιονομικές γραμμές που θα χρηματοδοτούν την κυβερνοασφάλεια. Απλώς θέλουμε ένα καλύτερο ορισμό και να έχουμε καλύτερη αντίληψη των συγκεκριμένων δαπανών αλλά και του αντικτύπου που έχουν για να πιάνουν τόπο τα κονδύλια αυτά. Δεν έχουμε ούτε καλό σύστημα δικτών, ούτε ποσοτικοποίηση για να έχουμε μια σαφή αντίληψη των δαπανών και των αποτελεσμάτων τους. Τώρα σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς και θα ολοκληρώσω με αυτό το θέμα γιατί ο κύριος Θαρθαλέχος ρώτησε και για τους οργανισμούς οι οργανισμοί έχουν δεδομένες αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, η ΕΝΙΣΑ, ο ΕΝΙΣΑ, ο Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, προτάθηκε να είναι ο συντονιστής, ε, ο συντονιστικός φορέας της Ένωσης για τις ε, κυβερνοεπιθέσεις. Αλλά τα κράτη-μέλη προτίμησαν τελικά να διατηρήσουν αυτά την αρμοδιότητα για τέτοια ζητήματα. Και η ΕΝΙΣΑ να διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο. Πάντως διαπιστώνουμε ότι οι οργανισμοί αυτοί, ο ΕΝΙΣΑ, η Europol, ο ΣΕΡΤΟ έχουν προβλήματα προσωπικού, δεν έχουν αρκετά καταρτισμένους υπαλλήλου. Ε, γιατί είναι δύσκολο να προσελκύσουμε και να κρατήσουμε ταλέντα. Υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα. Άλλωστε, ε, οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν κυρίως με προσωρινό αποσπασμένο προσωπικό από τα κράτη-μέλη. Και υπάρχει μεγάλη εναλλαγή, περιτροπή. Είναι δύσκολο λοιπόν να κρατήσουμε αυτά τα ταλέντα στους οργανισμούς, ε, ενώ αυτό θα χρειαζόμασταν. Αυτά και ολοκληρώνω. Μα τελειώνει ο χρόνο και έχουμε ακόμα άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αν έχετε όμω κάτι επιπρόσθετο να απαντήσετε, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σα, αν είναι αυτό δυνατόν. Να συμπληρώσω το εξή. Γι' αυτό πρώτο ο κ. Μπράιερ. Μιλήσατε για κάποιες από τις ενημερώσεις που έχουν γίνει από τότε που δημοσιεύτηκε η, ενημέρωση. Η ασφάλεια προφανώς είναι ένας τομέας που εσύ εξελίσσεται διαρκώς, κοιτώντας όμως το σύστημα πιστοποίηση, Βλέπουμε ότι υπάρχει δουλειά ακόμα να γίνει για να είναι αποτελεσματική. Αυτό που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την ασφάλεια αποτελούν ε, τα βασικά στοιχεία για την ε, συμμόρφωση. Και επίσης έχουμε και την ε, οδηγία για την ασφάλεια δικτύων. Αν ρωτάτε λοιπόν κατά πόσον υποστηρίζουμε την επισήμανση προϊόντων, δεν θα τοποθετηθούμε Κοιτάμε το θέμα της λογοδοσίας, της ευθύνη των παραγωγών και των προμηθευτών α, λογισμικού και υπηρεσιών σε ό,τι αφορά επίσης ε, και το θέμα της σωστής ε, φροντίδας των προϊόντων. Για το τελευταίο θέμα, το θέμα της διατήρησης δεδομένων. Εμείς το εξετάσαμε από την εξής οπτική γωνία. Κοιτάξαμε τι συνέπειε τη συνοριακή συνεργασία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πιστεύουμε ότι έχουμε να καλύψουμε κενά στο νομοθετικό πλαίσιο, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια σε ό,τι αφορά τις σωστές ε, έρευνες στον τομέα του κυβερνού εγκλήματο. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικό στι δηλώσει μου. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρονικό όριο. Είδε τον ημερωτικό έγγραφο για την προετοιμασία της έκθεσης ε, οδήγησε σε πολλές ερωτήσεις και πολλά σχόλια. Αυτό ενδεχομένως ε, να αποτελεί ένα δείγμα ότι θα πρέπει να σας ε, ακούσουμε ξανά στο μέλλον για πιο πολλές λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ήταν πολύ ωφέλιμη μεταλλαγή απόψεων και καλή επιτυχία σας εύχομαι στη δουλειά σας. Συνάδελφοι, τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Δημιουργία εργαλείου χρηματοδοτικού για την διαχείριση των ε, σύνορων. Η συγγητρία μας, η κυρία Φαγιών, είναι εδώ, η οποία θα μας πει τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που έχουν λάβει η χώρα. Ευχαριστώ πολύ και Τάνια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφοι. Να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο, για τις διαπραγματεύσεις που διεξαγάγονται για το εργαλείο για τη διαχείριση συνόρων και τις θεωρήσεις. Υπό τη Φιλανδική Προεδρία έχουν διοργανωθεί δύο τριμερείς ε, διάλογοι, προγραμματίζεται και ένας τρίτος στα τέλη του έτους. Εκτός αυτού έχουμε τέσσερις τεχνικές συναντήσεις, οι οποίες είναι ακόμα υπό εξέλιξη. Υπήρξε κάποια πρόοδος αρχικά, ωστόσο έχω να πω ότι όλα τα πολιτικά συντήματα εξακολουθούν να είναι εκκρεμή. Γιατί έχουμε μόνο μερική δέσμευση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, συγγνώμη. Και το πιο βασικό θέμα, το μέγεθος του Ταμείου παραμένει ανοιχτό. Και το θέμα του συνολικού οικονομικού πλασίου είναι στο πεδίο διαπραγμάτευση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο το έχω προειδοποιήσει συχνά ότι θα πρέπει όλα τα στοιχεία να εγκριθούν σε κανονική νομοθετική διαδικασία προκειμένου να έχουν ίσα δικαιώματα και οι δύο νομοθέτε. Δεν είναι δυνατόν εμεί ως Κοινοβούλιο να μην μπορούμε να αποφανθούμε για την κλίμακα του μέσου και να πρέπει να πούμε μόνο ναι όταν συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν μας αγχώνει. Δεν έχουμε ακόμα λοιπόν το συνολικό φάκελο ακόμα και έχουμε μόνο μερική εντολή από πλευρά του Συμβουλίου. Συζητάμε λοιπόν πολύ γενικά τα αριθμητικά στοιχεία και αυτό προφανώς δεν είναι παραγωγικό. Πέραν τούτου, Έχουμε και κάποια εγκάρσια πολιτικά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε το καθένα ξεχωριστά, γιατί έχουν αντίκτυπο σε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα στον τομέα των ιστορικών υποθέσεων. Έχει διοργανωθεί και έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα μια οριζόντια τεχνική συνεδρίαση για να εξετάσει ακριβώ τα θέματα αυτά. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ζητούν ε, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα. Το Κοινοβούλιο, από την άλλη, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιε εγγύσει. Δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή στα κρατημέλη και στην ε, Επιτροπή για το πώ θα δαπανηθούν οι πόροι αυτοί. Γιατί όταν θα εγκριθεί ο κανονισμό αυτό, ε, θα καθορίσει το νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα 7 χρόνια. Άρα πρέπει να τα ορίσουμε σωστά όλα αυτά. Τώρα είναι η στιγμή λοιπόν να καθορίσουμε του όρου. Τώρα, να εξετάσουμε εν συντομία τέσσερι ε, βασικού ε, τομεί όπου έχουμε διαφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Καταρχά, για την χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τι τρίτε χώρε. Εδώ, εν γέννη, ο σκοπό χρηματοδότηση σε τρίτε χώρε ε, μέσω του εργαλείου αυτού είναι κάτι που αμφισβητούμε. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο έχει σκοπό τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων. Εσωτερικό εργαλείο, όχι εξωτερικό. Και αυτό το τονίζουμε σε διάφορες περιστάσεις, γιατί έχουμε άλλα εργαλεία για την εξωτερική δράση. Αυτά έχουν εφαρμογή σε άλλες χώρες και είναι πολύ πιο υψηλά σε πόσο από ότι αυτό το εργαλείο. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να περιορίσουμε μέσω του εργαλείου αυτού σε 4% τη χρηματοδότηση σε άλλες χώρες και για τις ε, θεματικές ευκολύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Συμβούλιο και Επιτροπή διαφωνούν με οποιοδήποτε όριο, δεν θέλουν να μπει οποιοδήποτε όριο στις δαπάνες αυτές. Εδώ λοιπόν συζητάμε το κατά πόσο θα υπάρχουν ποσοστά και τι ποσοστά θα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ένα ελάχιστο ποσοστό για κάποιο ε, συγκεκριμένο στόχο για την κοινή πολιτική για τη θεώρηση. Έχουμε δύο συγκεκριμένου στόχου, τη διαχείριση συνόρων και την κοινή πολιτική για τι θεωρήσει. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι και οι δύο στόχοι αυτοί θα χρηματοδοτηθούν επαρκώς. Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Και η κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντική με την διαχείριση των συνόρων και την αποτροπή του εγκλήματο. Πιστεύουμε λοιπόν από πλευρά του Κοινοβουλίου ότι τουλάχιστον 20% τη χρηματοδότηση θα πρέπει να δαπανηθεί για το σκοπό τη κοινή ε, πολιτική για τι θεωρήσει. Η αντίδραση και του Συμβουλίου και τη Επιτροπή είναι μάλλον ε, αρνητική. Ωστόσο, για μα ω Κοινοβούλιο αποτελεί βασικό θέμα. Τρίτο θέμα. Τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών υποχρεώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει διαβούλευση με διάφορες υπηρεσίες πέρα από τη Frontex, η Ιουλίζα και το, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα προσθέθηκαν στον κατάλογο των υπηρεσιών με τις οποίες θα γίνουν διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων. Επίσης, ενισχύσαμε με τις διατάξεις για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις σχετικές διατάξεις όταν εφαρμόζουν τα μέσα αυτά και σε ό,τι αφορά την εποπτεία και την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων. Σεβόμενη φυσικά την αρχή της ε, μη ε, επιστροφής. Ε. Και εδώ βλέπουμε κάποια βελεξία από πλευρά της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Συνεχίζουμε λοιπόν τις συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Το τέταρτο βασικό στοιχείο, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εδώ είναι σαφέστατο ο στόχο μα. Θέλουμε να ενισχύσουμε το κείμενο του κανονισμού το διδακτικό σε ό,τι αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αρχή της μη διάκρισης. Έχουμε ένα νέο άρθρο ειδικά για το θέμα αυτό και κάποια, κάποιες θεολογικές σκέψεις τις οποίες έχουμε προτείνει από πλευρά μα προς το σκοπό αυτό και εδώ πιστεύω ότι ενδεχομένως να πετύχουμε κάποια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πετύχουμε σύντομα ένα σεμιβασμό ικανοποιητικό για τα θέματα αυτά, αλλά Κλείνοντα, θέλω να τονίσω εκ νέου ότι η τελική συμφωνία του κειμένου θα είναι μόνο δυνατή εφόσον το Συμβούλιο συμφωνήσει για το σύνολο του πολιτικού δημοσιακού πλαισίου, το οποίο δεν το περιμένουμε πριν από την επόμενη άνοιξη. Και στη φάση αυτή οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο φαίνονται πιο δύσκολες, γιατί οι δύο πλευρές ε, εμένουν στις θέσεις τους αλλά αυτό δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τις ομάδες διαπραγμάτευσης για την υποστήριξή τους. Πολύ ωφέλιμες ως τώρα. Και τους εισηγητές και τους συμβούλους στη Φιλανδική Προεδρία που προσπάθησε να περάσει μια πιο επικοδομητική προσέγγιση, αλλά όπως σας είπα μια και δεν έχουμε το τελευταίο, τελευταίο φάκελο, το νηστικό φάκελο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τι λεπτομέρειε. Ευχαριστούμε, Τανιά. Και ξέρουμε και ότι οι τρει τομεί, η διαχείριση συνορών, οι θεωρήσει, αλλά και το θέμα των οικονομικών ε, προκοποτήσεων είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα έχουμε και τα θέματα τη εντολή, τα οποία περιπλέκουν ακόμα την κατάσταση. Αλλά βλέπω ότι έχουμε μαζί μα και τουλάχιστον έναν σκιώδη εισηγητή να δώσω το λόγο στον κύριο Πίτερσε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι λακωνικότατο. Ήθελα να ευχαριστήσω την Τάνια Φαγιόν, την εισηγήτρια, για την εργό προσπάθεια στο θέμα αυτό. Είχαμε τεχνικούς, ε, τεχνικές συζητήσεις και τριμερείς διαλόγους. Καλή λοιπόν η προσπάθεια της κυρίας Φαγιόν και του επιτελείου της ε, διατρανώνοντας τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια είναι μερική εντολή διαπραγμάτευση του Συμβουλίου, όπως μας είπε η κυρία Φαγιόν. Εξού και η περιορισμένη πρόοδος που επιτυχάνεται. Δεν θα επαναλάβω τα όσα μας ανέφερε η συγγήτρια για μια αποτελεσματική